Okay, και κύριοι συνάδελφοι, όσοι εξημών είστε εδώ, να καθίσετε για να αρχίσουμε τη συνεδρίαση. Καλημέρα σε όλους και όλους. Να αρχίσουμε με την έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Αν δεν έχετε σχόλια καλά, να αρχίσουμε να προχωρήσουμε μάλλον στις ανακοινώσεις της Προέδρου όπου θα ήθελα πρώτα να θέσω υπόψη σας τη σύσταση των συντονιστών να αναδειχθεί ως εισηγήτρια η κυρία Μετσόλα για τέσσερις εκθέσεις για την συμμετοχή στο Asylum Support Office των, της Ελβετίας, Λίχτενστάιν, Νορβηγίας. Έχετε καμιά Ένσταση όχι. Καλά λοιπόν. Δεύτερο, δεύτερη ανακοίνωση της, Προέδρου, της Προέδρου. Προφορική ερώτηση για την ε, πολιτική προξενικών θεωρήσεων με γραπτή διαδικασία στις 22 Ιανουαρίου όπου οι συντονιστές αποφάσισαν να προωθήσουν προφορική ερώτηση στην Κομισιόν για την πολιτική προξενικών θεωρήσεων και αυτή να υποβληθεί το συντομότερο δυνατόν στην ε, Ολομέλεια. Αυτό λοιπόν πρέπει να, ε, για να γίνει αυτό πρέπει να εγκριθεί σήμερα. Δεν έχετε ενστάσεις. Και τέλος, για, τις, ε, για την διερμηνία. Δεν θα υπάρχουν φιλανδικά, εστονικά, μαλτέζικα και κροατικά το πρωί, το δε απόγευμα δεν θα έχουμε δανέζικα, φιλανδικά, τσέχικα, λετονικά και μαλτέζικα πάλι λόγω του περιορισμένου αριθμού των θαλαμίσκων διερμηνίας. Φαίνεται να μας κόβουν γλώσσες αρκετά τακτικά. Τώρα, υποτίθεται θα προχωρήσουμε στην παριθμόν 3. Αλλά ο εισηγητής ή η εισηγήτρια κυρία Γκαμπριέλ δεν είναι ακόμα εδώ. Ας προχωρήσουμε λοιπόν κατευθείαν στο τροποποίηση της αποφάσεως 2005-681 για την ίδρυση της ΣΕΠΟΛ, Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, με εισηγήτρια την κυρία Κίνγκα Γκάλ. Σήμερα συζητούμε την νομοθετική πρωτοβουλία 25 χωρών μελών για να πάει από το Μπράμσιλ στο Ενωμένο Βασίλειο η Αστυνομική Ακαδημία, η έδρα της δηλαδή στην Βουδαπέστη. Υπάρχει και χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο διότι η Βρετανική κυβέρνηση θα κλείσει μέχρι το καλοκαίρι την έδρα της ΣΕΠΟΛ. Άρα πρέπει να βρεθεί λύση πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Θα δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Γκάλ και μετά στους σκιώδεις εισηγητές, άλλα μέλη, Προεδρία του Συμβουλίου δηλαδή και Κομισιόν. Η κυρία Κίνγκα Γκάλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως και εσείς εξηγήσατε, η κατάσταση που διαμορφώνεται εδώ έχει ως εξής. Είναι σαφές ότι η ΣΕΠΟΛ, το όλο θέμα του οργανισμού αυτού δηλαδή, πρέπει να επιληθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, διότι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η ορθή λειτουργία του οργανισμού. και επομένως να λυθεί το πρόβλημα της έδρας το συντομότερο δυνατό. Όπως έχουμε πει εδώ στην παρούσα Επιτροπή και μάλιστα κατ' επανάληψη στο παρελθόν, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό ο οργανισμός που λειτουργεί ορθά και που ε, παίζει σημαντικό ρόλο να παραμείνει ανεξάρτητος. Για το λόγο αυτό υπάρχει ανάγκη να εξευρεθεί η κατάλληλη έδρα για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του. Είχαμε τώρα την πρωτοβουλία 25 χωρών μελών, όπως εξηγήσατε, και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που λύνεται το πρόβλημα με τον τρόπο αυτό, με την διαδικασία αυτή δηλαδή διατηρούνται, διαφυλάσσονται τα προνόμια του Κοινοβουλίου, είναι σαφής η διαδικασία ότι είναι συναπόφαση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως τόνισα ήδη, νομίζω ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο ανεξάρτητος χαρακτήρας και η ορθή λειτουργία του οργανισμού ΣΕΠΟΛ και άρα να βρεθεί η καλύτερη λύση το δυνατόν συντομότερο. Γι' αυτό άλλωστε περιέλαβα στο σχέδιο εκθέσεώς μου την σύσταση των 25 χωρών μελών η έδρα αυτή να εγκατασταθεί στην Βουδαπέστη. Υπάρχει και το θέμα τώρα του μέλλοντος της ΕΠΟΛ. Και αυτό το θέμα το θίγω στην σύντομη εκθεσή μου, γιατί είναι σαφές για όλες μας ότι η ΣΕΠΟΛ πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη συνθήκη λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, η ΣΕΠΟΛ πρέπει να παίξει κεντρικό ρόλο και μέσα στα νέα προγράμματα εκπαίδευσης για την επιβολή του νόμου και της τάξης Γι' αυτό περιλαμβάνω στο σχέδιο εκθέσεώς μου το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού ΠΟΛ που θα πρέπει να κατατεθεί σύντομα. Αυτά είναι λοιπόν τα σημαντικότερα σημεία της ε, σύντομης εκθεσής μου και είμαι διατεθειμένη να διαπραγματευτώ με τους και συγκητές για να βρούμε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπίσουμε και την πίεση χρόνου και να μπορέσει να ψηφιστεί η έκθεση πριν από την λήξη της θητείας μας. Η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών είναι η 4η Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Σκιώδης η κυρία Γκόνς από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Λίγα λόγια, διότι το έχουμε συζητήσει ήδη κατ' επανάληψη και η ομάδα μας συμφωνεί άλλωστε. Να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία της ΕΠΟΛΑ από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά συμφωνούμε ότι υπάρχει πίεση χρόνου διότι η νυν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο θα κλείσει, πρέπει να βρεθεί ένα καινούριο αρχηγείο της ΕΠΟΛ και γνωρίζουμε ότι και το Συμβούλιο συμφώνησε επί της Βουδαπέστης. Το ερώτημα είναι εάν μπορούμε να κλείσουμε τον φάκελο πριν από το τέλος της ε, θητείας. Συμφωνώ λοιπόν και με το χρονοδιάγραμμα που προτείνει η ε, Καγκάλ. Υπάρχει και προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Θα εξετάσουμε κάποιες τροπολογίες, αλλά ας προχωρήσουμε, ας προωθήσουμε ε, το θέμα αυτό για να τροποποιηθεί ο κανονισμός. Ευχαριστώ. Κύριος Δε Γιόγκ. Ευχαριστώ στα αγγλικά κύριε Πρόεδρε, καθώς και την εισηγήτρια για την ε, εξήγηση του θέματος. Με απογοητεύει λίγο ο τρόπος με τον οποίο ασχολούμεθα με το θέμα. Όλοι βέβαια συμφωνούμε επί της διαδικασίας, συναπόφαση, επ' αυτού δεν διαφωνώ, αλλά ανέμενα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφόσον συμμετέχει σε διαδικασία συναποφάσεω, να τα πάρει τα πράγματα σοβαρά υπόψη και να εξετάσει και κάποιε εναλλακτικέ επιλογέ. Δεν κατανοώ πολύ καλά γιατί η ΣΕΠΟΛ χρειάζεται να έχει βεβαίω ανεξάρτητη εντολή αλλά γιατί πρέπει να συμμορφωθούμε αμέσως με την σύσταση του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την έδρα ίσως να μην παρακολούθησα την ε, συζήτηση για τις εναλλακτικέ επιλογές εδώ στην Επιτροπή. Γιατί υπήρχαν και άλλες υποψήφιες χώρες. Εκτός από την Ουγγρική. Αν θέλουμε λοιπόν να πάρουμε στα σοβαρά το πράγμα και δεν νομίζω ότι εδώ πρέπει να μας εμποδίσει αυτή η πίεση χρόνου, διότι μπορούμε να αποφασίσουμε αρκετά σύντομα και επί εναλλακτικών επιλογών, αλλά δεν είδα να γίνεται η συζήτηση αυτή για εναλλακτικέ επιλογές και τώρα με σπρώχνουν να λάβω την απόφαση ότι δεν και καλά η Βουδαπέστη πρέπει να είναι η έδρα. Σε άλλη επιτροπή του ελέγχου του προϋπολογισμού προσπαθήσαμε, σταθήκαμε πολύ επικριτικά απέναντι σε έναν αριθμό οργανισμών και βεβαίως και με την έδρα των οργανισμών. Αν από τη μια μεριά έχετε λοιπόν την Ευρωπόλ, όπου συλλέγονται πολλές αστυνομικές πληροφορίες σε ένα μέρος και αλλού πλέον, τελείως αλλού, έχετε την ε, αστυνομική εκπαίδευση, νομίζω ότι αυτό δεν συμβαδίζει διόλου με τους στόχους τουλάχιστον της Επιτροπής Ελέγχου Προεπολογισμού. Λοιπόν, θα καταθέσω τροπολογίες για να κάνουμε τα πράγματα αυτά καλύτερα και όχι με τόση βιασύνη. Ευχαριστώ, De Jong. για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο. Εδώ έχω σημειώσει ένα όνομα, κυρίως η κυρία Σρεσέν. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε. Λουίτζι Σορέκα, τμήματάρχης ε, του τμήματο υπεύθυνου για την αστυνομική συνεργασία, σχέσει με την Europol και την Αστυνομική Ακαδημία. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω λίγο τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το θέμα αυτό. Θα γνωρίζετε ίσως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια γνωμοδότηση για την ε, ε, πρωτοβουλία των κρατών μελών στις 16 Ιανουαρίου η γνωμοδότηση αυτή αξιολογεί την πρωτοβουλία των κρατών μελών επί τη βάση τριών στοιχείων κατά βάση. Οι λειτουργικές συνέργειες που υπάρχουν ε, αφενός ως προς τη στήριξη και την αστυνομική συνεργασία, τα οποία διασφαλίζει η Europol, και αφετέρου το θέμα της ε, εκπαίδευσης ε, του αστυνομικού δυναμικού, που είναι το βασικό καθήκον της Αστυνομικής Ακαδημίας. Το δεύτερο κριτήριο ήταν η ευθυγράμμιση ε, των δαπανών ε, βάσει και της κοινή προσέγγισης ε, που έχουν εγκρίνει τα τρία θεσμικά όργανα για την αποκέντρωση και επίσης το τρίτο κριτήριο που κατά την άποψή μας είναι εξίσου σημαντική ότι η γνωμοδότηση έγινε βάσει της συνεχιζόμενης διαπραγμάτευσης μιας πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ε, τον κανονισμό της Ευρωπόλ, ο οποίος ακόμα είναι υποσυζήτηση στο Συμβούλιο και η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να προσθεθεί σε αυτή την, στην ε, πρωτοβουλία για την Αστυνομική Ακαδημία. Ακούσαμε ιδιαίτερα προσεκτικά το τελευταίο μήνα ε, και τα όσα μας έχουν πει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κρατημέλη στο Συμβούλιο που είναι κατά της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, στον κανονισμό της Europol ε, για τη συγχώνευση και επομένως κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε κάποιες εναλλακτικέ λύσεις για την πρόταση με στόχο να επιτύχουμε αυτό το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε κάποια στοιχεία στη γνωμοδότηση, όπως για παράδειγμα το να συστεγάζονται και τα δύο όργανα στη Χάγη. Και όπως είπε και η συγγήτρια ε, σήμερα, ούτως ή άλλως οι δύο οργανισμοί από και λειτουργικής σκοπιάς είναι ανεξάρτητοι. Υπάρχει μια τροποποίηση που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Είναι μια έκκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της ε, απόφασης του Συμβουλίου και να ευθαγραμμίσει τα πάντα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εδώ συμφωνούμε με τη θέση της εισηγήτριας. Θεωρούμε ότι το διάστημα των 18 μηνών αρκεί και από πολιτικής αλλά και από τεχνικής σκοπιάς μπορούμε να αξιολογήσουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να εξυγχρονίσουμε καλύτερα την Αστυνομική Ακαδημία. Όλα αυτά βέβαια ανάλογα και με τις αλλαγές που θα γίνουν στα θεσμικά όργανα αλλά είμαστε ευνοϊκά διακείμενοι και θεωρούμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πρόταση για να μπορέσουμε να ευθυγραμμίσουμε την Αστυνομική Ακαδημία με τη συνθήκη της Λισαβόνας εντός του χρονικού ορίου που μας ε, έθεσε η εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Η Ελληνική Προεδρία θέλει να λάβει το λόγο, να κάνει σχόλια. Δεν ξέρω ποιος είναι εδώ, παρακαλώ. Thank uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Από πλευρά Συμβουλίου και εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι το θέμα επήγει και πρέπει να υπάρχει και η βέλτιστη δυνατή λύση. Συνεδριάσαμε ήδη προκειμένου να εξετάσουμε το έγγραφο ε, της πρότασης των 25 κρατών μελών. Δεν έγινε κάποια αλλαγή στο σχέδιο κανονισμού. Εκτιμούμε το γεγονός ότι από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες και φυσικά βασιζόμαστε στη συνεργασία σας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει η απαραίτητη νομοθετική τροποποίηση εν ευθέτω χρόνο. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον όλων μας να συνεχίσει να λειτουργεί η Αστυνομική Ακαδημία και να μην είναι αβέβαια τα πράγματα για το προσωπικό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Um, then we come back to the Mrs. Ευχαριστώ. Ας, ας επιστρέψουμε τότε στην εισηγήτρια κυρία Κιν Γκαγκάλ. Άκουσα τις διάφορες απόψεις που εκφράστηκαν και θέλω να τονίσω και πάλι ότι νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την ορθή λειτουργία του οργανισμού. Διότι η δουλειά που κάνει είναι πολύ σημαντική και χρήσιμη. Και θα γίνει ακόμα πιο σημαντική. Και γι' αυτό προς το συμφέρον όλων μας δεν θα πρέπει να παρεμβληθούν εμπόδια. Γι' αυτό και εγώ ως εισηγήτρια θεωρώ επίσης ότι ο καλύτερος τρόπος για να διεξάγει το έργο του οργανισμός είναι να παραμείνει ανεξάρτητος και γι' αυτό νομίζω ότι η σύσταση που έχουμε και, που την έχω, και τα όσα έχω βάλει στην εκθεσή μου αποτελούν την καλύτερη εναλλακτική επιλογή για την ΣΕΠΟΛ. Βεβαίως είμαι ανοιχτή σε συζητήσεις με τους και οδησίτες Έχουμε προβλέψει και σχετικές συναντήσεις. Θα δούμε και τις τροπολογίες και θα επανέλθουμε στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Είπατε ότι μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου επειδή δεν έχει έρθει μέχρι τώρα ακόμη ο εισηγητής για, την προηγούμενη, για το προηγούμενο θέμα, το επόμενο θέμα της κυρίας Γκόνς Προβλέπετε στις 9.40, 40, δηλαδή σε λίγο περισσότερο από 10 λεπτά. Μήπως θέλετε να διακόψουμε για λίγο να προλάβουν να έρθουν όλοι. Μπορούμε να προχωρήσουμε, λέει η κυρία Κίνγκα Γκόνς. Μερικοί από τους κοιόδης ηγητές είναι, είναι παρόντες ή παρούσες. Και άρα μπορούμε να αρχίσουμε. Α, πολύ ωραία. Τότε να αρχίσουμε. Κλείστε το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ. Σημείο 5 λοιπόν οι σχέσει με την ε, ποινική δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Ε, στην ανακοίνωσή της για το πίνακα βαθμολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα νέο έγγραφο, μια ανακοίνωση που ε, επικεντρώνεται στη διοικητική δικαιοσύνη, αλλά ε, μας ενδιαφέρει κυρίως το ποινικό δίκαιο, η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου. Ε, η συζήτηση για το μηχανισμό για την διαφύλαξη του κράτους δικαίου εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόμα να εξελίξει και αναμένουμε ενδιαφέρουσες ε, προτάσεις στον τομέα αυτό. Να δώσω το λόγο λοιπόν στην εισηγήτρια, στην κυρία Γκόντς και κατόπιν να περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Προεδρία σε περίπτωση που θέλουν να λάβουν το λόγο και μετά θα γίνει συζήτηση μεταξύ των συναδέλφων. Παρακαλώ κυρία Γκέντς. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για ένα ακόμα πιεστικό ζήτημα, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει την ανακοίνωση για το θέμα αυτό στις αρχές Μαρτίου και θέλει να αποστείλει ένα πολύ στεναρό μήνυμα. Ελπίζει ότι θα υπάρξει ισχυρή πλειοψηφία στην ε, Επιτροπή μας. να υποστηρίξει τη θέση μας για το θέμα αυτό και να πω ότι η διαδικασία αυτή ξεκίνησε περίπου πριν από ένα χρόνο. Τον Απρίλιο εγκρίθηκε το θέμα αυτό από τους συντονιστές και ε, ήθελε το θέμα και Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ε, γιατί θεωρούσε ότι υπάρχουν θέματα αρμοδιότητας. Έγιναν κάποιες συναντήσεις με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και έτσι άλλαξε ο τίτλος και σταματήσαμε να μιλάμε για τον πίνακα βαθμολογίας και αναφέρεται ρητά το θέμα του ποινικού δικαίου και του κράτους δικαίου στον τίτλο και εξολόγηση της δικαιοσύνης. Μας εξέπληξε επίσης το γεγονός ότι όταν συμφωνήσαμε με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ότι είναι αρμοδιότητα της δικής μας της Επιτροπής και πάλι ε, θέλησαν να υποβάλουν γνωμοδότηση. Φαίνεται ότι λύθηκε βέβαια στο μεταξύ το ζήτημα διότι υπάρχει προθεσμία για την ε, ε γνωμοδότησή τους την επόμενη Δευτέρα και θα προλάβουν λοιπόν να μας τη δώσουν εγκαίρως πριν ε, την ε, ψηφοφορία στη δική μας την Επιτροπή. Έτσι ελπίζουμε να έχουμε τελειώσει τη ε, διαδικασία πριν το τέλος της αιτίας μας. Ήθελα απλώς να σας τα υπενθυμίσω όλα αυτά, διότι κάποιοι συνάδελφοι διαμαρτυρήθηκαν και είπαν ότι δεν υπάρχει χρόνος για να υποβληθούν τροπολογίες και να συζητηθούν συμβαστικές τροπολογίες, αλλά δεν είναι όλα χαμένα. Έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό από τον Απρίλιο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε ε, και το θέμα αυτό πριν το τέλος της θητείας. 73 τροπολογίες λάβαμε. Κάποιες από αυτούς προσθέτουν κάποια νέα στοιχεία στην πρότασή μας και αρχίσαμε πολύ νωρίς ε, να ε, ετοιμάζουμε συμβαστικές τροπολογίες για όλα τα θέματα. Εχθές συναντηθήκαμε με τους κοιόδης εισηγητές για να συζητήσουμε και αυτές τις συμβαστικές προτάσεις. Η έκθεση έχει τέσσερις βασικές προτάσεις. Πρώτον είναι ε, η επέκταση του ε, πίνακα βαθμολόγησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει και στοιχεία ποινικού δικαίου και μετά θα ασχοληθούμε ε, και με τη σχέση με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Υπάρχουν κάποιες συμβιβαστικέ τροπολογίες οι οποίες λένε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επεκταθεί ο πίνακας βαθμολογίας αλλά να υπάρχει ταυτόχρονα και έναν εξάρτητο μέσο αργότερα ίσως, το οποίο δεν θα έχει άμεση σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και ξέρουμε τώρα ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ήταν ο μόνος τρόπος να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Ελπίζουμε όμως ότι στην ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως μας υποσχέθηκαν, θα υπάρχουν και προτάσεις για πιθανές αλλαγές στο μέλλον. Και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε έναν εξάρτητο μέσο. Η άλλη βασική πρόταση είναι ότι ζητάμε ένα μηχανισμό για περιπτώσεις κρίσεως, ε, μια ταχεία αντίδραση και υπάρχουν αρκετές τροπολογίες που υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Επίσης ζητάμε ένα ε, καλό μηχανισμό αξιολόγησης, αυτό είναι πολύ σημαντικό και κάποιες από τις τροπολογίες ενισχύουν ακριβώς αυτή την άποψη. Και επίσης ε, έχουμε μια πολύ στενότερη συνεργασία και ε, θεσμική σχέση μεταξύ της Επιτροπής της Βενετίας και της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέλουμε να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, ζητά γνωμοδοτήσεις από την Επιτροπή της Βενετίας και φυσικά υπάρχει σχέση και μεταξύ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ε, περιγράφεται επίσης ο ρόλος και η σχέση με τα Εθνικά Κοινοβούλια σε κάποια παράγραφο του κειμένου. Ελπίζουμε να μπορέσουμε λοιπόν να εργαστούμε στο επόμενο διάστημα εντατικά και ζητώ και τη στήριξη των συναδέλφων για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό εγκαίρως, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει πίεση χρόνου. Έχουμε προγραμματίσει και μια συνεδρία την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο για να συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Βοηθήστε μας λοιπόν, σας παρακαλώ να το ολοκληρώσουμε αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γκέντς. Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει κάποιο ο οποίος θα ήθελε να σχολιάσει. Δεν έχει έρθει ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελληνική Προεδρία. No. Does any of the colleagues wish... Από του συναδέλφου, ο κύριο Δεγιάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ για να συμπληρώσω το κενό χρόνο, επειδή έχουμε πρόβλημα εδώ, ευπρόσδεκτη η έκθεση της King Agents. Νομίζω ότι και η σύνοψη που κάνατε για τα όσα συνέβησαν εχθέ και το πώς θα προχωρήσουν οι συμβαστικές τροπολογίες είναι καλή. Η βασική μου ανησυχία είναι ότι αν όλα αυτά τα θέσουμε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμένου, κατά πάσα πιθανότητα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα για την ανάγκη της αξιολόγησης της δικαιοσύνης. Βέβαια είναι οικονομικό αυτό το εξάμεινο που σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επισημάνεται την οικονομική αξία του νόμου και ορισμένες φορές μπορεί να υπάρχουν εντάσεις μεταξύ οικονομικών και δικαιοσύνης. Εμείς ε, προτιμούμε τη δικαιοσύνη, γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής ε, της ανακοίνωσης για να, ε, ανακοίνωσης για να περιλαμβάνονται και τα θέματα ποινικού δικαίου, όπως προτείνει η συγκήτρια, αλλά θέλουμε να έχουμε και ένα μηχανισμό ο οποίος εξετάζει όλες τις πτυχές και τις οικονομικές αλλά και τα θέματα της δικαιοσύνης, τις γενικότερες πτυχές της δικαιοσύνης. Γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε έναν ανεξάρτητο μηχανισμό, όπως είπε και η συγγήτρια. Αυτό κατά είναι το πιο σημαντικό θέμα και νομίζω ότι μπορούμε γρήγορα να ακολουθήσουμε την προσέγγιση που μας πρότεινε η συγγήτρια. Φυσικά θα συνεργαστούμε πλήρως για να βρεθούν συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ, κυρία Γκρίσπεκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω την εισηγητρία για το έργο της που το ολοκλήρωσε και γρήγορα. Εξαιτία και του χρόνου που ε, μεσολάβησε μεταξύ της απόφασης του Προεδρείου και της δυνατότητας να συζητήσουμε το θέμα στην Επιτροπή, έτσι ώστε να καταλήξουμε και στις συμβιβαστικές ε, τροπολογίες. Σε κάθε περίπτωση τον φάκελο αυτόν το κοινοβούλιο τον χειρίστηκε γρήγορα. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια. Δεν πήρα εγώ το λόγο για να συμπληρώσω το χρόνο όπως και ο συνάδελφος, αλλά για να πω ότι συμφωνούμε με την ανάγκη αξιολήγησης των δικαστικών συστημάτων όλων των κρατών μελών, κυρίως με βάση τις αρχές του κράτους δικαίου, τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις αξίες της, Ευρω... Ευρώπης. Και ταυτόχρονα πρέπει να το επιθυμίσουμε, όσο και αν φαίνεται τετριμένο, ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές ε, που θεμελιώνονται στον χάρτη σε όλα τα θεσμικά κείμενα. Κάτι που δεν συμβαίνει πάντα. Έχουν υποβληθεί μια σειρά τροπολογίες και κατά τη διάρκεια της συζήτησης τους και εκεί διαπιστώσαμε ότι η συγγήτρια κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Τρία σημεία εγώ θέλω να επισημάνω που είναι τα πιο σημαντικά κατά την άποψή μου και είναι αυτά που προσπάθησα να ε, ενισχύσω και μέσω των τροπολογιών μου. Πρώτα απ' όλα, αυτός ο πίνακας βαθμολόγησης δεν θα πρέπει να είναι απλώς ένα στατιστικό εργαλείο έτσι, με γραφικές παραστάσεις που να μας δείχνουν συγκριτικά τις διαδικασίες και τα λοιπά ενδιαφέρον έχουν, αυτό, έχουν αυτά αλλά το σημαντικό είναι να τα αξιοποιήσουμε για αξιολόγηση να αξιολογήσουμε τον τρόπο απονομή τη δικαιοσύνη, δηλαδή στα κράτη-μέλη. Όπως και ο συνάδελφο, με λυπεί το γεγονός ότι η Επιτροπή ε, βλέπει και θέτει αυτό το εργαλείο μόνο ως ένα οικονομικό εργαλείο στο πλαίσιο του εξαμήνου. Για χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο συζητάμε για την ανάγκη αξιολόγηση τη αποτελεσματικότητα των ε, συστημάτων απονομή δικαιοσύνη. Και μέσω αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε ένα εργαλείο για να την κάνουμε αυτή την αξιολόγηση. Και ιδιαίτερα την αξιολόγηση τη ε, ποινική δικαιοσύνη. Δεύτερο σημείο που θεωρώ σημαντικό, η προστασία και, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τα ίδια τα κράτη-μέλη, ακόμα ένα θέμα για το οποίο συζητάμε πολλά χρόνια τώρα, πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός από την Επιτροπή και αναφέρομαι στα λόγια του συναδέλφου πριν από λίγες εβδομάδες του Πλημισελ, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί αυτό το εργαλείο που θα παρακολουθεί το σεβασμό, αλλά ταυτόχρονα και μια διαδικασία που θα επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβιάσεων. Τρίτο θέμα, το οποίο προσπάθησα να εισάγω μέσω τροπολογίας γιατί δεν υπήρχε πουθενά. Πώς μπορεί να γίνει μια ολιστική, μια συνολική αξιολόγηση του συστήματος δικαιοσύνης όταν τα κράτη-μέλη αρνούνται να παράσχουν όλα τα στοιχεία. Τι θα κάνουμε δηλαδή σε περιπτώσεις που θα υπάρχουν κενά να που θα υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα του εργαλείου. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βρουν έναν κάπως εναρμονισμένο τρόπο να συλλέγουν τα ε, στοιχεία αυτά και κυρίως και σε κάθε περίπτωση να τα αποστέλουν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό προβλέπει το κείμενο. Αλλά επίσης και στα θεσμικά όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μόνο έτσι θα μπορεί να είναι αποτελεσματικό αυτό το εργαλείο και όχι απλώς μια συλλογή στοιχείων. Συμπερασματικά να πω ότι χαίρομαι για αυτό το, το αποτέλεσμα. Έχουμε ακόμα μια συνάντηση μπροστά μας και άλλη μία στο Στρασβούργο και ευελπιστώ ότι σύντομα θα συμφωνήσουμε και θα καταλήξουμε σε μια ε, ε, βαρύ ισχυρή ε, θέση από την πλευρά της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών για το θέμα αυτό. Αυτά είχα να πω από την πλευρά της πολιτικής μου ομάδας και πάλι ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ευχαριστούμε. Η Επιτροπή διαπιστώνω ότι ήρθε ο εκπρόσωπος της. Μήπως θέλετε το λόγο για το, την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθούμε από κοντά τις συζητήσεις στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών για την αξιολόγηση του συστήματος δικαιοσύνης και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτά όμως είναι δύο θέματα ξεχωριστά τα οποία δεν θα πρέπει να συγχέονται, κάτι το οποίο το αναδείξαμε ήδη από το Δεκέμβριο στη συζήτηση που είχαμε τότε και στην οποία πολλά μέλη της Επιτροπής εδώ συμμετείχαν. Με τον πίνακα βαθμολόγησης θα αξιολογούμε όλα τα ζητήματα που αφορούν στην απονομή της δικαιοσύνης, όχι μόνο το αστικό δίκαιο με τη στενή του έννοια. Και θεωρεί, γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή, ότι χρειάζεται χρόνος και δεν μπορούν να γίνουν τα πράγματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχουμε υποβάλει τροπολογίες, ή μάλλον θα καλωσορίζαμε τροπολογίες που θα μπορούσαν να υποβληθούν προς αυτή την κατεύθυνση ε, στην έκθεση. Το θέμα το ανέδειξε και ο πρόεδρος Ρόζο στην ε, ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης και προετοιμάζει μια ανακοίνωση η Επιτροπή ε, την Άνοιξη χρειάζεται να δημιουργηθεί μια διαδικασία επιβολής κυρώσεων στοχευμένη και πολιτική, από τη μια, ακόμα και μια διαδικασία η οποία θα προβλέπει την αναστολή ορισμένων δικαιωμάτων ε, κράτους, κράτους μέλους. Η εμπειρία μας είναι ότι η Επιτροπή έχει καταφέρει να λειτουργήσει ως ένας ε, ανεξάρτητος και ε, αντικειμενικός διαιτητής σε τέτοιου τύπου ε, διενέξεις. Οποτεδήποτε υπάρχει σοβαρό και συστηματικός κίνδυνος του ε, σεβασμού του κράτους δικαίου, τότε χρειάζεται ε, δράση. Κάποιες από τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί το αναφέρουν ότι χρειάζεται λοιπόν να δημιουργηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός και διαδικασία ταχεία επέμβαση σε περίπτωση κρίση. Δηλαδή σε περιπτώσει όπου υπάρχουν συστηματικές παραβιάσει ε, του κράτου δικαίου. Πράγμα που ταιριάζει με τη θέση που εξέφρασε και ο πρόεδρο Μπαρόζο. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα μηχανισμό έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοιε σοβαρέ καταστάσει και με τρόπο νόμιμο αλλά και σεβόμενη την ισότητα των κρατών μελών. Ευχαριστούμε η συγκήτρια θέλει να τοποθετηθεί. κλείνοντα τη συζήτηση, ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ και του συναδέλφου. Και τον εκπρόσωπο τη Επιτροπής. Τι διαπιστώνω από τις παρατηρήσεις που άκουσα, πάνω κάτω συμφωνούμε. Με όλα εκείνα που είπε ο πρόεδρος Παρόζο στην ε, ομιλία του, το έργο που έχει διεξάγει η Επιτροπή μας. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο μηχανισμό, ένα μηχανισμό αποτελεσματικό που θα είναι ε, αξιόπιτος, τόσο αντικειμενικός, θα βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά. Και κάτι ακόμα προσπαθούμε να τονίσουμε μέσω αυτή της έκθεσης και χαίρομαι και ευχαριστώ τους συναδέλφους που έχουν συμφωνήσει και έχουμε καταφέρει να εργαστούμε τόσο ε, γρήγορα. Και χαίρομαι επίσης που και η Επιτροπή συμφωνεί. Βέβαια όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είχαν συζητηθεί επί μακρόν παλιότερα. Νομίζω το μάθαμε το μάθημα εδώ στο Κοινοβούλιο και γενικότερα ότι χρειάζεται χρόνος για κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν σταδιακά, δεν μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό το έχουμε αποδεχθεί. Αλλά είναι σε κάθε περίπτωση σημαντικό να τα δημιουργήσουμε αυτά τα, αυτούς τους μηχανισμούς και αυτά τα εργαλεία. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, διαπιστώνω ότι η κυρία Γκάμπριελ δεν είναι παρούσα, επομένως θα ε, σταματήσουμε τη συνεδρίαση μέχρι τις 10 για να ξεκινήσουμε τότε τη ψηφοφορία.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 Colleagues, can I ask everybody... Η πρόεδρος κυρία Ιντφέλτ. Σας παρακαλώ καθίστε για να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Colleagues, please take your seats. Η πρόεδρος, κύριε Εντφέλη, σας παρακαλώ καθίστε για να αρχίσουμε. Colleagues, colleagues, uh, I would like to start the vote, but... Uh, θα ήθελα να αρχίσουμε. Βλέπω όμως ακόμη να καταφθάνουν διάφοροι από πολιτικές ομάδες. Έτσι, για δύο λεπτά θα παρακαλέσω την κυρία Γκάμπριελ να μας ενημερώσει για τις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται για την αναθεώρηση του 539 για την λίστα χωρών των οποίων οι πήκοοι απαιτείται να διαθέτουν προξενική θεώρηση για να εισέλθουν στον χώρο Σέγγεν. Κύριε Γκάμπριελ, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, για τον φάκελο που έχουμε ήδη ψηφίσει στις 21 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο. Λίγα προκατακτικά σχόλια πρώτα. Γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροποποίησε το κείμενο που αρχικά είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μεταφορά στον θετικό κατάλογο 16 χωρών, νησιωτικών χωρών ΑΚΕ με τέσσερις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, μία για την συμπερίληψη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Περού Κολομβία. Εκτός από την ομάδα αυτή των χωρών έχουμε εγκρίνει άλλες δύο τροπολογίες. Η πρώτη τροπολογία είναι σχετικά με το γεγονός ότι θέλουμε να εντάξουμε κριτήρια στην βάση των οποίων γίνεται η μεταφορά μέσα σε ένα άρθρο και όχι σε εκτιμώντας, σε αιτιολογική σκέψη δηλαδή. Επίσης αναφέρεται το Κοινοβούλιο στα θεμελιώδη δικαιώματα. Με άλλη τροπολογία δε αναφέρεται στο δικαίωμα να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τις υποεξέλιξη ε, διαπραγματεύσεις. Ο πρώτος τριμερής διάλογος έγινε στις 8 Ιανουαρίου. Αναμείναμε το Συμβούλιο να συμφωνήσει, να τεθεί επιτάπητος το θέμα. Ο πρώτος τριμερής διάλογος είδε, ε, ε, επέτρεψε να γίνει ένας καρποφόρος διάλογος και μετά προχωρήσαμε στις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε συμβιβασμό. Έγινε και δεύτερος τριμερής διάλογος, τούτην εδώ την εβδομάδα, στις 28 Ιανουαρίου. Βρισκόμαστε ακόμη στο στάδιο των συζητήσεων, τις οποίες συνεχίζουμε σε αναζήτηση συμβιβασμού. Είναι αναγκαίο τώρα να συνεχίσουμε να αναζητούμε λύσεις που να εξυπηρετούν και τα τρία θεσμικά όργανα, ιδίω βέβαια τους δύο συνομοθέτες, Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Τώρα ακόμα δύο θέματα συμφωνήσαμε για την συμπερίληψη Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Περού και Κολομβίας. Σε ό,τι αφορά Κολομβία και Περού, η μεταφορά θα γίνει μετά από αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αξιολόγηση αυτή θα διαβιβαστεί, θα κοινοποιηθεί δηλαδή και στο Κοινοβούλιο. Το δεύτερο, όπως είπα πριν, αναφέρεται στην τροπολογία που προτείνει τα κριτήρια να ενταχθούν σε άρθρο του ίδιου του κανονισμού, ακόμα δεν έχουμε καταληξεί συμβιβασμό, και το τρίτο για την υποχρέωση δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενημερώνει το Κοινοβούλιο. Εκεί σε καλό δρόμο βρισκόμαστε για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Τώρα βρισκόμαστε στην φάση διατυπώσεως νέων τροπολογιών για να μπορέσουμε να έχουμε έναν τρίτο τριμερή διάλογο την επόμενη εβδομάδα στην περίοδο συνόδου του Στρασβούργου. Εκεί βρίσκεται λοιπόν το θέμα. Ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους και όλους και ήθελα απλώς να ενημερώσω τους συναδέλφους και σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία. Ευχαριστώ κυρία Γκαμπριέλ, λέει η πρόεδρος Σιντφέλτ. Νομίζω τώρα όλοι έχετε σαφή εικόνα της διαδικασίας και ας αρχίσουμε με την πρώτη ψηφοφορία στο θέμα 6 της ημερήσιας διάταξης για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ευρωπόλ και την κατάργηση των κανονισμών 681 και 0091 με εισηγητή τον κύριο Αγουστίν Δίας Έχετε, θέλετε να γράψετε το λόγο κύριε εισηγητά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μια πολύ σύντομη παρέμβαση για να ευχαριστήσω εξαιρετικά για το έργο τους ε, και για τη γενναιόδορη βοήθειά τους όλους τους ε, σκιώδεις εισηγητές και όλους όσους υπέβαλαν τροπολογίες. Νομίζω ότι καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό παρά το γεγονός ότι υπάρχει διάσταση πολιτικών απόψεων και σήμερα θα καταφέρουμε να αποστείλουμε ένα μήνυμα συνένεση, συνένεση για τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ και πάλι εκ βάθους καρδίας. Σας ευχαριστώ. Προχωρούμε τώρα στην ψηφοφορία. Πρώτη ψηφοφορία είναι για το σύνολο τροπολογιών. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τώρα τροπολογία 23 του εισηγητού υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Θέλετε επαλήθευση. Καλά. Προχωρούμε σε ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τροπολογία 23. Ψηφίσατε. Λήξεις. Απερίφθη λοιπόν, όντως. Ή 23 πάντα, έτσι. 23. Ψηφίσατε μόλις την τροπολογία 23. Απερίφθη. 194 τώρα υπέρ, κατά, απορρίπτεται και αυτή. Τροπολογία 25 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 205 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 206 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται. ...205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θα ήθελα όμως να επαναληφθεί. 215, συγγνώμη, 215 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται αυτή. Κάποιες εκπίπτουν. Οι τροπολογίες 29 και 30 μαζί, υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογίες 2, 224, 2, 24 και 26 όλες μαζί υπέρ, κατά. Θα ήθελα επαλήθευση παρακαλώ. Νομίζω ότι εγκρίνονται. 222, 22, 24, 26. Ψηφίσατε. Λήξη. Απορρίπτονται λόγω ισοψηφία. Ε. Καλά κάναμε και παρέθεσαμε. 223. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2.25. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 227 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά εγκρίνεται 231 υπέρ κατά εγκρίνεται 33 α με ναι αυτή εκπίπτει 232 υπέρ κατά απορρίπτεται 2.33 υπέρ κατά απορρίπτεται 34 υπέρ κατά εγκρίνεται. 2.34 υπέρ κατά εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά εγκρίνεται. 36 και 37 μαζί υπέρ κατά εγκρίνονται. 235 με προφορική τροπολογία του εισηγητού να εγκριθεί δηλαδή ως 10α υπέρ κατά εγκρίνεται 38 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 39 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 40 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 2.36 υπέρ, κατά απορρίπτεται, 2.37 υπέρ, κατά εγκρίνεται, συμβαστική 8 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 242 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά εγκρίνεται και αυτή. 2.45 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά εγκρίνεται 251 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική 11 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά εγκρίνεται 43 το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται, αλλά ας επαληθεύσουμε. Δεύτερο τμήμα τη 43. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Δείξει. Εγκρίνεται τελικά. Η επόμενη εκπίπτει, εκπίπτει, εκπίπτει. 13, συμβαστική 13. Υπέρ κατά εγκρίνεται 46 υπέρ κατά εγκρίνεται 47 υπέρ κατά εγκρίνεται 48 υπέρ κατά απορρίπτεται 49 υπέρ κατά εγκρίνεται 264 υπέρ κατά εγκρίνεται. 265 υπέρ. Με συγχωρείτε, εκπίπτει αυτή. 50 υπέρ. Υπέρ. 50. Κατά. Απορρίπτεται. 266 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 268 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 267 υπέρ κατά απορρίπτεται 269 υπέρ κατά απορρίπτεται 270 υπέρ κατά απορρίπτεται και αυτή 271 με προφορική όπως ε, η προηγούμενη υπέρ κατά εγκρίνεται 51 υπέρ κατά εγκρίνεται 52 υπέρ κατά απορρίπτεται 272 υπέρ κατά εγκρίνεται 273 υπέρ κατά εγκρίνεται επαλήθευση καλά 273 ψηφίσατε λήξη Εγκρίνεται λέει η πρόεδρος, αλλά προφανώς κάνει λάθος. Απορρίπτεται, απορρίπτεται. Δεν βλέπω, δεν <laughs> φαίνεται καλά την οθόνη μου, ναι. Η 56 τώρα υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 282, 312 και 314, όλες μαζί υπέρ, κατά. Είναι πολύ κοντά η πλειοψηφία και η μεψηφία Ας γίνει επαλήθευση. Ψηφίσατε. Λήξη. Εγκρίνεται λοιπόν. Πράγματι. Παρακαλώ να σηκώνετε καλά τα χέρια γιατί αλλιώ θα χρειαστεί να κάνουμε διαρκώς επαληθεύσεις. 57 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 283 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Κοντ 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2, 87, 88, 301, 2, Όλες μαζί υπέρ κατά εγκρίνονται. 289 υπέρ κατά εγκρίνεται. Θέλετε επαλήθευση. 289 λοιπόν η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε. Λήξη. Α, ήταν όλες μαζί. Νόμιζα ότι είχατε όλοι μπροστά σας τη, τη λίστα ψηφοφορία και ήταν σαφές για σας. Πάντως εγκρίνεται τώρα. Προχωρώ στη συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Κοντ 6 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Επαλήθευση. Καλώς. Κοντ 6. Εάν ψηφίσατε όλες και όλοι, τότε λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 296, 297, 317 υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 67 έχει αποσυρθεί. 298 υπέρ, κατά, Απορρίπτεται νομίζω, αλλά ας επαληθεύσουμε. Ψηφίσατε. Λήξη. Εγκρίνεται. Παρακαλώ και πάλι να σηκώνετε καλά τα χέρια. Διότι αν από κάθε ομάδα σηκώνει ένας δυο τα χέρια, τι να κάνω, είμαι υποχρεωμένη να μαντέψω. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται 69 υπέρ κατά εγκρίνεται 308 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 18 υπέρ κατά εγκρίνεται 309 υπέρ κατά εγκρίνεται 71 υπέρ κατά εγκρίνεται 19, συμβαστική δηλαδή 19 υπέρ κατά εγκρίνεται 73 του εισηγητού υπέρ κατά εγκρίνεται 74 υπέρ κατά εγκρίνεται κοντ 7 υπέρ κατά εγκρίνεται 75 υπέρ κατά εγκρίνεται όλες μαζί τις 55-77 μέχρι κάτω-κάτω 147 μέχρι την 147 υπέρ κατά εγκρίνονται α εκπίπτει αυτή συμβαστική 20 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβαστική 21 υπέρ κατά εγκρίνεται 3.44 υπέρ. Εγκρίνεται. 3.55 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 3.64 και 65 υπέρ. Κατά εγκρίνονται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 380 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 381 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 382 υπέρ. Κατά. Ε, απορρίπτεται νομίζω. Αλλά ας κάνουμε παρήθευση. 382. Ψηφίσατε. Λήξη. 42 προς 7 βεβαίως. Εγκρίνεται. Αρκετά σίγουρα. Συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τέσσερα μηδέν πέντε υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Α, μάλλον εκπίπτει αυτή. 26 συμβαστική υπέρ κατά εγκρίνεται και καλύπτει πολλές. Α, υπάρχει κάποια τροπολογία ενδιάμεσα. 406 υπέρ. Δεν είμαι βέβαια για τις τεχνικές λεπτομέρειες, πάντως φαίνεται ότι πρέπει να ψηφίσουν 406 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας επαληθεύσουμε. Ψηφίσατε. Λήξη. Εγκρίνεται λοιπόν πράγματι. Και κάνουμε ένα μεγάλο άλμα. 4.41 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 4.42 και 43 υπέρ κατά εγκρίνονται 444 υπέρ κατά εγκρίνεται 445 6 αυτές οι δύο υπέρ κατά απορρίπτονται θέλετε επαλήθευση Κατά. 445 και 46 Λήξη. Απερίφθησαν λοιπόν. 4.47 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα 4.63, 64, 65, 66 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 467, 68, 69 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 471 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται ομοίως. 470, 72, 73 υπέρ. Κατά. Αυτές μάλλον οι μόνοι 473 έτσι. Εγκρίνεται. Εκπίπτουν ορισμένες. 476, 77, 78 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 479 και 81 υπέρ κατά εγκρίνονται ψηφίζεται ως προσθήκη 480 υπέρ κατά απορρίπτεται αυτή εδώ 482 θέλετε επαλήθευση επαλήθευση 480 λήξη εγκρίνεται 482 υπέρ κατά απορρίπτεται 483 υπέρ κατά εγκρίνεται 486 υπέρ κατά εκπίπτει λέει η πρόεδρος α η επόμενη 487 υπέρ κατά απορρίπτεται 491 υπέρ κατά εγκρίνεται 493 και 95 ταυτόσημες υπέρ κατά απορρίπτονται επαλήθευση καλώς 493 και 95 εγκρίνονται. 4,96 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 4,97 και 500 ταυτόσημες υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. 4,98 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 501 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 502 και 504 ταυτόσιμες υπέρ κατά εγκρίνονται. 505 υπέρ κατά εγκρίνεται. 506 και 7 υπέρ κατά απορρίπτονται. 513 υπέρ κατά εγκρίνεται μετά εκπίπτουν 2.509 υπέρ κατά εγκρίνεται 511 υπέρ κατά εγκρίνεται 514 υπέρ κατά εγκρίνεται 516 υπέρ κατά εγκρίνεται 5 όχι 5 5.17 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτή. 5.15 εκπίπτει. 5.18 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5.19 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 5-20 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 521 υπέρ. Κατά απορρίπτεται, νομίζω. 522 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 524 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 525 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 526 27 υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 528 υπέρ, κατά απορρίπτεται 529 υπέρ κατά εγκρίνεται 531 υπέρ κατά εγκρίνεται 532 υπέρ κατά εγκρίνεται 534 και 35 μαζί υπέρ κατά εγκρίνονται 536 υπέρ κατά απορρίπτεται 37 υπέρ κατά απορρίπτεται 538 υπέρ κατά εγκρίνεται 540 540 υπέρ κατά εγκρίνεται και αυτή 542 υπέρ κατά απορρίπτεται 544 υπέρ κατά Εγκρίνεται. 5.46. Θέλετε επαλήθευση. Ωραία. Κάνουμε επαλήθευση λοιπόν την 5.44. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 5.46 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 5.47 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 5.48 υπέρ κατά, εγκρίνεται, 5.50 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 5.53 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 5.55-5.56 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 5.57-58 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 5.59 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 560 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 562 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 563 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 564 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, Συμβαστική τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 5,76, εβδομήντα Βάιντεν Χόλσερ υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 586, 299, 313 μαζί υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. Ε, επαλήθευση. Ψηφίζουμε τις 586, 299 και 313 μπλοκ. Άρχεται ψηφοφορία, πέρασες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 5.95 υπέρ. Α, είναι προσθήκη. Ψηφίζουμε την 5.85 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται ως προσθήκη. Η 5.85 ήταν αυτή. Ωραία. 5.95 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 5.97 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 101 προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται, αλλά θα ήθελα να κάνουμε μια επανλήθευση, Ψηφίζουμε την 101 ως προσθήκη. Μία ψήφος επιπλέον. Ψήφισαν όλοι. Ωραία, πέραση της ψηφοφορια εγκρινεται Εγκρίνεται, όντως. 610-611 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 613 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 6-17 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 6-19 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 6-21 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 31 υπέρ. Συμβαστική τροπολογία 31. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την 635 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 32 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 113 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, κόντα 11 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 644-645 υπέρ, επαλήθευση για την κόντα 11. Επαλήθευση της κόντα 11 λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ωραία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 644-645 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Κοντ 12 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Κοντ 13 και 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνονται. Αύκο 27 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Κοντ 14 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Επαλήθευση για την 116 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 663 υπέρ κατά απορρίπτεται απορρίπτεται θέλετε να κάνουμε επαλήθευση εντάξει επαλήθευση για την 663 της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 664 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 665 με προφορική τροπολογία από το συνεισηγητή που προσθέτει το Especially Women and Children υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 666 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 667 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Και περνάμε σε αιτιολογικές σκέψεις. 127 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Αύκο 3 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 134 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά απορρίπτεται 137 υπέρ, κατά εγκρίνεται 140 υπέρ, κατά απορρίπτεται 141 υπέρ, κατά απορρίπτεται 138 υπέρ, κατά απορρίπτεται 139 υπέρ, κατά εγκρίνεται τροπολογία 9 υπέρ, Υπέρ. Υπέρ. Ωραία. Κατά. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Κόντα 1 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 149 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 150 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 151 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 152 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 15 από τον εισηγητή υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Κοντ 2 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 154 και 156 υπέρ, κατά, εγκρίνονται. 18 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 160 υπέρ, κατά απορρίπτεται, 162 υπέρ, κατά απορρίπτεται, 161 υπέρ, κατά απορρίπτεται, 163 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 165 υπέρ, κατά εγκρίνεται, 166 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά. Δεν ε, μπορώ να δω. Σηκώστε τα χέρια σας. 169 υπέρ. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Ε, κατά. Εγκρίνεται. 171 υπέρ κατά εγκρίνεται. 172 υπέρ κατά εγκρίνεται. 173 υπέρ κατά εγκρίνεται. 174 υπέρ κατά εγκρίνεται. 175 υπέρ κατά εγκρίνεται. 176 υπέρ κατά εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά εγκρίνεται. 180 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 183 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 186 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 187 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Αύκο 7 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 188 υπέρ κατά εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα τώρα, budget 1 υπέρ κατά εγκρίνεται. Budget 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. Budget 3 υπέρ κατά. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά να το επαληθεύσουμε. Η τρία της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Ψήφισαν όλοι. Λείπει μία ψήφος. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Budget 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Και φτάνουμε στο τέλος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Μπράβο σας. Περνάμε λοιπόν στην επόμενη ψηφοφορία για την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας ε, ε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Μέλλο είναι εισηγητής. Θέλετε το λόγο. Ωραία λοιπόν, περνάμε απευθείας στην ψηφοφορία. Συγχαρητήρια στον κύριο Διάστητε Μέρα και πάλι. Τώρα όμως έχουμε να ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Μέλο. Συμβαστική τροπολογία α, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 που μπορεί να ε, ψηφιστεί ως προσθήκη στη συμβαστική α, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, Κατά. Απορρίπτεται. Επαλήθευση για την τροπολογία 3. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται, είχατε δίκιο. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά, εγκρίνεται, τροπολογία 7 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, τροπολογία 8 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, τροπολογία 9 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, τροπολογία 10 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, τροπολογία 11 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 12 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 13 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά εγκρίνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν ε, ηλεκτρονικά το σύνολο του κειμένου. Άρχεται η ψηφοφορία. Δύο ψήφοι ακόμα. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορία. Εγκρίνεται με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Η ίδια με την προηγούμενη έκθεση. Συγχαρητήρια στον κύριο Μέλο. Και περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία για σήμερα. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάπτυξη του συστήματος e-call σε οχήματα και ε, τροποποιώντας την ε, ε, οδηγία 2007-46. Ο συντάκτης της νομοδότησης είναι ο κύριος Βος. Θέλετε το λόγο κύριε Βος. Δεν θέλετε το λόγο. Ωραία. Ψηφίζουμε. Υπολογία 19. η οποία ψηφίζεται μαζί με την 27, 31, 34, 39, 41, 44 και 50 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20, η οποία συνδέεται με διάφορε άλλε τροπολογίε που βλέπετε στον κατάλογό σα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 44. Επίση ψηφίζεται μαζί με διάφορε άλλε. Υπέρ. Κατά. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 45. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 47, ζητώ συγγνώμη, 46, η οποία ε, συνδέεται με διάφορες άλλες, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 49 υπέρ, Κατά. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 53. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 54. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Εδώ έχουμε τμήματική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. Έχει αποσυρθεί η 6. Καταπίπτουν διάφορες μια και συμβαστική 2. Και ψηφίζουμε για την ε, περίεργη αυτή η ψηφοφορία, λέει η Πρόεδρος. «80 και μετά ε, θα επανέλθουμε στην 77». Ένα λεπτό, ένα λεπτό να λύσουμε τη γραμματεία. Okay. We go to Ωραία, 80. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται, αλλά ας ελέγξουμε. Νομίζω ότι εγκρίνεται, ας ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας για την 80 πρώτο τμήμα. υπέρ ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα λοιπόν καταπίπτει. Νομίζω. 87 λοιπόν υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται στι ιδεολογικέ σκέψει. 21 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 24 και 25 μαζί υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 1 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 27 υπέρ. Όχι, ζητώ συγγνώμη. Καταπίπτουν διάφορε και πηγαίνω 31 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 32 έχει καταπέσει. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Βλέπετε. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 43 3 υπέρ. Απορρίπτεται. Είχε καταπέσει 43 λοιπόν. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά, έναρξη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Συγχαρητήρια. Και ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες για σήμερα. Συνάδελφοι, πρέπει να διακόψουμε, γιατί είχε προβληθεί ότι το επόμενο θέμα θα ξεκινήσει στις 11.30 και η Επιτροπή δεν έχει έρθει ακόμα, ο πρόσωπός της, επομένως διακόπτουμε στις 11.30.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 Uh, colleagues, shall um, Συνάδελφοι, ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Έχουμε μια κοινή συζήτηση για τα σημεία 9 και 10 από κοινού που αφορούν στι συμφωνίε Ευρωπαϊκή Ένωση Αζερβαϊτζάν, αφενό για την επανεισδοχή προσώπου που διαμένουν χωρί άδεια και αφετέρου για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. Συγγετρία είμαι η κυρία Κάπριελ και για τις δύο από το ΕΛΚ. Πρόκειται για διαδικασία συγκατάθεσης. ήθιστε οι συμφωνίες επανεισδοχής να εγκρίνονται μαζί με συμφωνίες απλούστευσης έκδοσης ε, θεωρήσεων, ξενικών θεωρήσεων. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην εισηγήτρια και μετά στην Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για το γεγονό ότι βρίσκεται εδώ, γιατί ε, προσωπικά προετοιμάζω το προσχέδιο της έκθεσης που θα παρουσιαστεί στις 12 και 13 Φεβρουαρίου. Και χαίρομαι λοιπόν που η Επιτροπή έχει έρθει εδώ και θα μπορέσει να μας δώσει μερικές πληροφορίες περισσότερες για τις δύο αυτές συμφωνίες που εξετάζει η Επιτροπή μας. Πρώτα λοιπόν θα ήθελα να ακούσω την άποψη της Επιτροπής για να έχουμε περισσότερε πληροφορίε για το που βρίσκονται οι διαπραγματεύσει. Πώ έχουν διεξαχθεί αυτέ οι διαπραγματεύσει. Και μετά εγώ θα ήθελα να ξαναλάβω το λόγο για να απαντήσω σε αυτέ τι πληροφορίε. Ωραία. Άρα πρώτα δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή, λέει η πρόεδρο. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Με χαρά να σας ενημερώσουμε για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2012 Είχαμε τέσσερις συναντήσεις διαδοχικές για τις δύο αυτές τις ε, συμφωνίες και διάφορες ανεπίσημες συναντήσεις επίσης και καταφέραμε τελικά τον Ιούλιο του 2003 να συμφωνήσουμε. Για τις εκτός θεωρήσεων υπογράφτηκε η σχετική συμφωνία τον Νοέμβριο και αναμένουμε σύντομα την υπογραφή της ε, συμφωνίας για την επανεισδοχή προσώπων. Αναμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου που θα εξουσιοδοτεί αυτή την υπογραφή. Φυσικά δεν μπορεί να αρχίσει να ισχύει, να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία για την Απλούστευση εκτό Θεωρήσεων χωρί ταυτόχρονα να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία επανεισδοχής στον αφορά την επανεισδοχή μπορώ να σας ενημερώσω ότι είναι η συνηθισμένη συμφωνία η οποία καλύπτει όλα τα στους υπηκός τρίτων χωρών και όλες οι υποχρεώσεις του, της τρίτης χώρας ε, ως ήθιστε είναι αμοιβέ. Καταγράφονται επίσης λεπτομερώς οι διαδικασίες για την επανεισδοχή και οι σχετικές προθεσμίες. Υπάρχουν προβλέψεις επίσης και για τους ε, ταξιδιώτες ε, που ε, διέρχονται, transit, καθώς επίσης και για επιταχυμένες διαδικασίες στα σύνορα. Θεωρούμε ότι κυρίως αυτή η συμφωνία θα αφορά υπηκός Αζερμπαϊτζάν, επανεισδοχή υπηκών Αζερβαϊτζάν, μιας και δεν έρχονται από τη χώρα αυτή για λόγους γεωγραφικής θέσης, πολύ υπηκόοι τρίτων χωρών. ούτε έχουμε διαπιστώσει μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα να περνούν από το Αζερβαϊτζάν. Να χρησιμοποιούν τη χώρα αυτή ως χώρα τράνζιτ. Και τρίτον, οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις μάλλον για την επανεισδοχή υπηκών τρίωτων χωρών είναι πολύ συγκεκριμένες και αφορούν σε περιπτώσεις μόνο ε, α, που, που, που το πρόσωπο έχει αμέσως αφιχθεί στο Αζερβαϊτζάν, άρα μόνο δια της αεροπορικής οδού. Η επανεισδοχή είναι προς τη χώρα προέλευσης και όχι προς τη χώρα τράνζιτ, η οποία θα ήταν το Αζερβαϊτζάν στην περίπτωση αυτή. Θα ήθελα να ευστήσω την προσοχή σας σε κάποιες νέες προβλέψεις οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί και έχουν σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι οποίες συμπεριλήφθηκαν μετά από την ε, σημαντική αναθεώρηση, ανασκόπηση των συμφωνιών απανεσδοχής που ανέλαβε η Επιτροπή. Και κυρίως αναφέρομαι στο άρθρο 2 για τις θεμελιώδεις αρχές. Ένα παρόμοιο άρθρο συμπεριλήφθηκε στη Συμφωνία Επανεισδοχής με την Αρμενία που υπογράψαμε πρόσφατα και αυτό προβλέψει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσώπων ε, που τίθενται σε διαδικασία επανεισδοχής θα πρέπει να γίνονται σεβαστά και αυτό ισχύει και σε περιπτώσεις εθελούσιας επιστροφής και σε απελάσεις, αναγκαστικές επιστροφές. Και καταγράφεται στο σκήμενο της συμφωνίας ότι όλες, όλο το σχετικό διεθνές δίκαιο, όπως για παράδειγμα η Συμφωνία της Γενέβης για το δίκαιο των προσφύγων, και ο θεμελιώδης κάτω ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Προβλέπεται επίσης μια ρήτρα η οποία μπορεί να ε, ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που διαπιστωθεί σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερβαϊτζάν. Μια και εδώ δεν έχουμε πολλές, ε, ε, πολλή μετανάστευση από τρίτες χώρες, εδώ δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρχει μεγάλος αντίκτυπος αυτής της ρήτρας. Πρόκειται λοιπόν για διαδικασία συγκατάθεση. Ε, θα δώσω το λόγο στη συνάδελφη να σα δώσω περισσότερε λεπτομέρειε για την ε, Συμφωνία Απλούστευση εκτό θεωρήσεων. Ευχαριστώ τον συνάδελφο. Όπω εξήγησε, πάντα συμφωνούμε, ε, μάλλον διαπραγματευόμαστε σαν πακέτο από κοινού τέτοιου τύπου συμφωνίε, δηλαδή επανεισδοχή και απλούστευση βίζα. Οι διαπραγματεύσεις αυτές γίνανε στο πλαίσιο της ε, ανατολικής ε, γειτονίας, ε, εταιρικής σχέσης μάλλον, που προβλέπουν την σύναψη τέτοιων συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Έχουμε ήδη ενισχύ τέτοιες συμφωνίες με τη Γεωργία, με την Ουκρανία, με τη Μολδαβία και την Αρμενία δηλαδή περισσότερες από τις χώρες της ε, Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Η μόνη η οποία δεν ε, συμπεριλαμβάνεται είναι η Λευκορωσία. Αλλά με την ευκαιρία μπορώ να σας ενημερώσω ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσουμε ε, διαπραγματεύσεις και με τη Λευκορωσία. Αυτή η συμφωνία απλούστευσης θεωρήσεων είναι πολύ παρόμοια με εκείνη που συνάψαμε με την Αρμενία. Σε γενικέ γραμμές καλύπτει τις ίδιες κατηγορίες προσώπων οι ίδιοι ταξιδιώτες θα υποφελούνται από τις προβλέψεις της, υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ αυτής της συμφωνίας και της συμφωνίας με την Αρμενία. Εδώ πρόκειται για συμφωνία όπου υπάρχει πλήρης αμοιβαιότητα. Μιας και το Αζερβαϊτζάν είχε ακόμα ε, την απέτηση οι υπηκοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκδίδουν προξενική θεώρηση. Το οποίο σημαίνει ότι αυτή η νέα συμφωνία θα αλλάξει το καθεστώς βίζας που χρειάζεται για τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταξιδεύουν προς το Αζερβαϊτζάν. Είναι κάπως τυποποιημένες οι διατάξεις. Ε, μειώνεται ο χρόνος που χρειάζεται για την επεξεργασία και την έκδοση της προξενικής θεώρησης. Σύμφωνα με το συνήθι ε, κώδικα για τις προξενικές θεωρήσεις είναι 15 ημέρες. Μειώνεται επίσης το τέλος, αντί για 60 ευρώ σε 35 ευρώ και για ορισμένες κατηγορίες ταξιδιωτών μάλιστα απαλλάσσονται πλήρως από το, την υποχρέωση καταβολής αυτού του τέλους. Υπάρχουν και άλλες ε, συνήθεις διευκολύνσεις για διάφορες κατηγορίες Για παράδειγμα, ε, χρειάζεται, δεν χρειάζεται να υποβάλουν τόσο πολλά δικαιολογητικά που να εξηγούν το σκοπό του ταξιδιού. Και κάτι σημαντικό, ε, θα δίνεται η δυνατότητα να εκδίδονται πολλαπλέ θεωρήσει, θεωρήσει πολλαπλή εισόδου, σύμφωνα με το άρθρο 5. Και τέλος, κάτι που επίσης συνηθίζεται ε, προβλέπεται το γεγονό ότι δεν θα χρειάζονται τα διπλωματικά ε, διαβατήρια, οι κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρίων να εκδίδουν προξενική θεώρηση. Θα διαπιστώσετε στο τέλος ότι υπάρχει μια κοινή δήλωση για τα υπηρεσιακά διαβατήρια. Το Ζερβαϊτζάν ήθελε να υπάρξει απαλλαγή προξενικής θεώρησης και για τα υπηρεσιακά διαβατήρια, όμως εμείς δεν είχαμε τέτοια εντολή και γι' αυτό δεν συμπεριλήφθησαν τα υπηρεσιακά διαβατήρια στη συμφωνία. αλλά τόσο πολύ του ενδιέφερε το Αζερβαϊτζάν να έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει διμερείς διαπραγματεύσεις ε, προς αυτή την κατεύθυνση με τα κράτη-μέλη, που συμφωνήσαμε να συμπεριληφθεί στο τέλο τη συμφωνία μια κοινή δήλωση, η οποία λέει ότι τίποτα από αυτά που αναφέρονται στη συμφωνία δεν ε, αποκλείει τη δυνατότητα του Αζερβαϊτζάν να κινήσει διεμερείς διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη για τα υπηρεσιακά διαβατήρια. Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία. Όπως είπε και ο συνάδελφος, καλωσορίζουμε την έκθεση της ε, εισηγήτριας και φυσικά θα απαντήσω οποιαδήποτε ερώτημα έχετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι κανείς εδώ από πλευράς Ελληνικής Προεδρίας. Ωραία. Να πάμε πρώτα στην εισηγήτρια τότε και έχει ζητήσει και κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο. Κύριε Γκαμπριέλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς ε, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας ε, έκανε μια διεξοδική παρουσίαση και μας παρουσίασε τη σημασία αυτής της έκθεσης ε, και τις σχέσεις. Πρόκειται για εμβάθυνση και προώθηση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αζερβαϊτζάν στα πλαίσια βέβαια της ανατολικής εταιρικής σχέσης και φυσικά ε, πρόκειται και για μια πολύ σημαντική ε, διαδικαστική ε, διευκόλυνση και βλέπουμε ότι απλουστεύουμε και επιταχύνουμε αρκετές διαδικασίες. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας υπενθύμησε ότι πρόκειται για δύο συμφωνίε οι οποίες δεν μπορούν να τεθούν σε ισχύ παρά μόνο ταυτόχρονα. Ε, η διαδικασία είναι μια διαδικασία έγκρισης και θα ήθελα επίσης να επιμείνω και σε κάποια ε, σημεία. Καταρχάς, ε, την αρχή της αναλογικότητας. Υπάρχει και το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, το οποίο αναφέρεται ρητά στην έκθεση για την επανιστοχή. Ε, και θεωρώ ότι χάρη σε αυτές τις δύο εκθέσεις ε, μπορούμε να εκφράσουμε την πολιτική μας υποστήριξη για να ενισχύσουμε την κινητικότητα σε περιβάλλον ασφάλειας. Για μας λοιπόν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Θα ήθελα επίσης να σταθώ και ε, στο θέμα της έκδοσης προξενικών θεωρήσεων. Θα γίνονται όλα πιο γρήγορα, μειώνονται τα τέλη Ίσως όμως και μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, αν θα υπάρχουν ε, διάφορες ε, περιπτώσεις εφαρμογής για διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κάποια κράτη για τα οποία δεν θα ισχύει αυτό το καθεστώς. Ε, καλό θα ήταν να μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες εδώ στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Και όσον αφορά την έκθεση για την επανεισδοχή, μας χαροποιεί το γεγονός ότι υπάρχουν όλα τα τεχνικά στοιχεία, ότι υπάρχει μια πιο ταχεία διαδικασία και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η συμφωνία προβλέπει και τη δημιουργία μιας μικτής επιτροπής επανεισδοχής η οποία θα φροντίζει να εφαρμόζεται σωστά η συμφωνία ε, και ε, θα ήθελα να ξέρω πώς θα μπορούσαμε να λάβουμε περισσότερο υπόψη το ρόλο του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτές είναι οι πρώτες ερωτήσεις που έχω να θέσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διεξοδική παρουσίαση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι οι εκθέσεις αυτές αδιαμφισβήτητα αποτελούν πρόοδο στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε στη συνέχεια το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει τις ερωτήσεις. Η κυρία Κρίσπερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Καταρχάς να καλωσορίσω μία ομάδα δημάρχων από τη Γαλλία και να τους πω ότι δεν θα πρέπει να πιστέψουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μόνο γυναίκες, γιατί σήμερα έχουμε μόνο γυναίκες ευρωβουλευτές εδώ στην αίθουσα. Ε, καμιά φορά έχουμε και κανέναν άντρα. Μην ε, σας ε, ε η σημερινή εικόνα. Να ευχαριστήσω λοιπόν τώρα την κυρία Γκαμπριέλ για το έργο της, το οποίο ξεκινάει τώρα και την ευχαριστώ επίσης που πρότεινε πριν παρουσιάσει καν την έκθεσή της να δώσει το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα διότι ε, βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο της συμφωνίας που έπρεπε να μας δώσει πληροφορίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, πριν από κάποιες μέρες είχαμε την αντίστοιχη παρουσίαση για την ε, Τουρκία. Δεν ήταν τόσο καλή η ισορροπία και να ευχαριστήσω επίσης διότι λαμβάνουμε υπόψη και τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και του Αζερβαϊτζάν μέσω αυτών των δύο συμφωνιών. Και μας ενδιαφέρει ο διάλογος, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός ε, και μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών της ε, σχέσης Ανατολικής Γειτονίας και αυτές τις συμφωνίες σύνδεσης που συνάπτονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, με την Αρμενία, τη Μολδαβία. Όλες αυτές ε, θα πρέπει να ε, ολοκληρωθούν μέχρι και τη Λευκορωθουσία. Όλες αυτές οι χώρες λοιπόν της Ανατολικής Γειτονίας ή έχουν προσπογράψει τις συμφωνίες αυτές ή είναι στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και είναι στα πρόθυρα της υπογραφής και θεωρώ ότι αυτές είναι πάρα πολύ θετικές πολιτικές ενδείξεις για τις χώρες αυτές, διότι και από την πλευρά τους και από τη δική μας υπάρχει μια περιφερειακή λογική η οποία συνεισφέρει στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις ε, χώρες του Νοτιού Καυκάσου. Και Ελπίζω, ε, αυτό βεβαίως προφανώς το επιθυμούμε όλοι, αλλά ελπίζω ότι όντως ε, θα ε, διευκολύνουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ανάπτυξη του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και φυσικά των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά φυσικά και με τα δικαιώματα του ανθρώπου όλες τις κατάλληλες εξελίξεις για να υπάρχει ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες αυτές. Δεν έχω πολλά σχόλια να κάνω για τη συμφωνία ε, για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων διαβατηρίων. Ε, μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις διάφορες περιπτώσεις, τη δυνατότητα προσορμαγής ε, όσο το δυνατόν καλύτερα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όλοι γνωρίζουν ότι η διευκόλυνση προξενικών θεωρήσεων είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη και για τους ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τις χώρες αυτές, αλλά και για μας στην ε, γυραιά Ευρώπη που έχουμε ανάγκη να μην ε, είμαστε μία ήπειρος η οποία ε, θα γίνει σύμφωνα με την διατύπωση του Γκίφερ Φερχόφστατ το... η ε, γυράσκουσα κοινωνία. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια καλή σχέση μεταξύ των ε, ε, παλιών και των νέων και όλων αυτών των χωρών. Θα ήθελα λοιπόν να υπενθυμίσω αυτή την ανησυχία που την έχω συνεχώς για όλες αυτές τις συμφωνίες διότι αυθόρμητα θέλουμε να δώσουμε την ε, σύμφωνη γνώμη μας για τους ε, ανθρώπους, ε, τους πολίτες του Αζερβαϊτζάν, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο πάντα μου δημιουργεί πρόβλημα. Από ό,τι θυμάμαι υπάρχει η συμφωνία με το Πακιστάν, την οποία δεν είχα βρει ικανοποιητική και ελπίζω να μην είμαι και η μόνη διότι είχα θεωρήσει ότι δεν είχαμε παρκείς ε, πληροφορίες και δεν υπήρχε κατάλληλη αξιολόγηση της κατάστασης για τους ανθρώπους αυτούς που κατάγονται από αυτή τη χώρα ε, για... και οι οποίοι θέλουν να έρθουν στα ευρωπαϊκά εδάφη. Όσον αφορά το Αζερβαϊτζάν, η χώρα έχει υπογράψει τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Ε, εδώ λοιπόν έχουμε ούτως ή άλλως μια πολύ ισχυρή εγγύηση, έχει προσυπογράψει και την Σύμβαση των ε, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά γνωρίζουμε ότι τα πρόσφατα γεγονότα στο Ζερβαϊτζάν, πιο συγκεκριμένα ε, η σύγκρουση και με, ε, για την περίπτωση του Ναγκόρνο Καραμπάχ με την Αρμενία, μπορεί να μας δημιουργήσει κάποιες ανησυχίες και φυσικά από εκεί προέρχεται και η δική μου ανησυχία. Για να ολοκληρώσω με δύο λόγια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως υπενθυμίσατε και εσείς κυρία μου, και πολλές φορές εγώ έχω ρωτήσει τη Σεσίλια Μάλστρομ ε, εάν πρέπει να γίνει κατάλληλη αξιολόγηση και παρακολούθηση για τους ανθρώπους αυτούς, τους οποίους επιστρέφουμε στις χώρες τους. Πρόκειται για πολύ ευάλωτες δημοκρατίες η Επίτροπος είχε δεσμευθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενώπιον της Επιτροπής μας να μας δώσει πληροφορίες για το πώς εφαρμόζονται αυτές οι συμφωνίες επανεισδοχής. Εσείς μας είχατε παρουσιάσει την κατάσταση, μας υπενθυμίσατε και την αξιολόγηση η οποία είχε γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011, αλλά εγώ θα ήθελα ε, πολύ πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και να μην έχουμε απλώς ε, μια χρονολογική σειρά των ε, περιστάσεων, ε, όχι για το τι υπογράφεται. Τις συμφωνίες τις γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Μας ενδιαφέρει η πρακτική εφαρμογή των συμφωνιών αυτών, πόσους ανθρώπους αφορούν, ε, τι γίνεται με την πανένωση οικογενειών, αν ε, στέλνουμε πίσω οικογένειες που έχουν και μικρά παιδιά. Λίγα πράγματα για την κατάσταση αυτών των ανθρώπων που στέλνουμε στις χώρες τους από τα ευρωπαϊκά εδάφη. Και φυσικά υποστηρίζω απόλυτα την τελευταία παράγραφο της αιτιολογικής έκθεσης της ε, εισηγήτριας, χρειαζόμαστε να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή της ε, συμφωνίας και μας ενδιαφέρει η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, χαίρομαι ιδιαίτερα για το περιεχόμενο ε, της έκθεσης της συναδέλφης μου που προεδρεύει σήμερα, τη Σόφι ε, για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και στην ανάγκη για διαφάνεια για όλα αυτά τα θέματα. Ε, με συγχωρείτε που μακρηγόρησα, είχαμε και χρόνο σήμερα γιατί δεν έχουμε και πάρα πολλούς βουλευτές στην αίθουσα. Ευχαριστώ. Thank you. Um, can the commission brief... Ευχαριστώ. Η Κομισιόν μπορεί να απαντήσει σύντομα στις ερωτήσεις της εισηγητρίας. Μία σύντομη ερώτηση της εισηγήτριας για την ε, διευκόλυνση της έκδοσης προξενικών θεωρήσεων, συμφωνία αυτή δηλαδή, εφαρμόζεται σε όλους, καλύπτει όλους τους υπηκός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός όσων δεν, δεν συμμετέχουν στο χώρο του Σέγγεν, δηλαδή Δανία, Ιρλανδία και Ενωμένο Βασίλειο. Για τις χώρες αυτές προσαρτάται στο τέλος της συμφωνίας κοινή δήλωση που λέει ότι οι δοθήσεις της ειδική θέσεώς των εκφράζεται η επιθυμία να συνάψουν παρόμοιες συμφωνίες με το Αζερβαϊτζάν οι χώρες αυτές. Ευχαριστώ. Εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Πρώτα για την Συμφωνία Επανεισδοχής. Την, για την μεικτή Επιτροπή Επανεισδοχής. Αυτή έχει ήδη συνδεθεί και θεσπιστεί. Είναι σημαντικό όργανο παρακολούθησης. Στην Επιτροπή αυτή εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τις χώρες μέλη. Συμμετέχουν βεβαίως και οι ομόλογοι μας από την πλευρά των Αζερμπαϊτζανών. Είναι κυρίως ο υδραυλικός η Επιτροπή αυτή, δηλαδή συζητεί τα καθημερινά θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της συμφωνίας. Κάθε φορά που μια χώρα μέλος αντιμετωπίζει ένα εμπόδιο στην καθημερινή εφαρμογή μπορεί να το θέσει στα πλαίσια της ε, Επιτροπής αυτής, η οποία προσφέρει την ε, πλατφόρμα για να εξευρεθούν λύσεις. Υπάρχει εκεί η δυνατότητα να προσκληθούν και τα τρίτα μέρη, κάτι το οποίο γίνεται με κοινή συνένεση των δύο μερών και σύμφωνα με τους ε, κανόνες εσωτερικών διαδικασιών. Επίση η ερώτηση της βουλευτού σας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι αυτό έχει θεμελιώδη σημασία και σε σχέση με τη συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν αλλά και γενικότερα για όλη την πολιτική επανεισδοχής. Επανέρχομαι στα προηγούμενα σχόλια μου, αν με επιτρέπετε, για την επανεισδοχή τρίτων, τρίτων χωρών και απάτριδων δεν μπορούμε να του βάλουμε συμφωνία αυτή για τους λόγους που εξήγησα προηγουμένω και που έχουν σχέση με, με τις πολύ περιοριστικές συνθήκες ή, ή μάλλον όρους που περιλαμβάνει η μαλλον ορους Επανεισδοχής. Επίσης, το κεκτημένο ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Return Directive εφαρμόζονται πλήρως. Δεν επιτρέπει καταστατήγηση των διατάξεων αυτών η Συμφωνία Επανεισδοχής Εάν κάποιος κινδυνεύει με την επιστροφή του στο Αζερβαϊτζάν, δεν μπορεί να επιστραφεί στο Αζερβαϊτζάν. Είτε υπάρχει συμφωνία επανεισδοχής ή όχι, η οποία έχει απλώς διοικητικό χαρακτήρα και μπορεί να επιστραφεί. Αυτή είναι η νομική πραγματικότητα. Η συμφωνία επιμένει για να διασφαλίσει ότι τα πράγματα είναι έτσι, περιλαμβάνει και διασφαλίσεις και η αξιότιμη βουλευτής τόνισε ότι το Αζερβαϊτζάν έχει συνυπογράψει όλες τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Η σημασία του λεγόμενου post-return monitoring, παρακολούθηση μετά την επιστροφή δηλαδή, είναι επίσης σημαντική. Μετά από τις συζητήσεις με το Κοινοβούλιο για το Πακιστάν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε σκληρά για να ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει αυτή την παρακολούθηση μετά την επιστροφή για την Ουκρανία και το Πακιστάν. Έχει αρχίσει η διαδικασία αυτή. Συνεργαζόμαστε και με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης καθώς και με τον ύπατο αρμοστή για τους πρόσφυγες των Ενωμένων Εθνών και το πρόγραμμα αυτό θα διαρκέσει τρία έτη και αναμένουμε από αυτό το πρόγραμμα να μας προσφέρει πολλά χρήσιμα δεδομένα όχι μόνο όσον αφορά την ευμερία των επιστρεφωμένων προσώπων Ουκρανία και Πακιστάν αλλά και γενικότερα για την δυνατότητα εφαρμογής αυτού του post-return monitoring που είναι δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία και γι' αυτό ακριβώς το πιλωτικό πρόγραμμα θα μας επιτρέψει να εξαγάγουμε συμπεράσματα. Και μετά από την τριετία αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι σε θέση να καθορίσει εάν αυτό το post-return monitoring μπορεί να εφαρμοστεί και σε ευρύτερη κλίμακα. Αρκούμε σε αυτά. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος Ιντφέλτ. Κυρία Συγκίτρια. Άλλο, τίποτα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μια ερώτηση. Αφού πρώτα ευχαριστήσω και τη συναδελφό μου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πληροφορίες που μας διέθεσαν και τις επισημάνσεις που έκαναν, που είναι σημαντικά δηλαδή για την μελλοντική έκθεση και εγώ ως εισηγήτρια σημειώνω τις πληροφορίες αυτές για να μπορέσω να τις θέσω υπόψη των συναδέλφων μου με διαρθρωμένο τρόπο. Απλώς λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω για μια φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τακτικό διάλογο και για το θετικό πνεύμα συνεργασίας που έχει επιδείξει και που ελπίζω να συνεχίσει να επιδεικνύει. Σας ευχαριστώ, λέει η πρόεδρος Σόφια Ιντεφέλντ και τώρα... Είναι κάπως ε, δρόμος μετεμποδίων, διότι έχουμε φτάσει ακριβώς στο μεσημέρι, αλλά δεν βλέπω πουθενά τον εισηγητή. Α, έρχεται μου λέτε. Ελπίζω να είναι όντως τουλάχιστον μέσα στο κτίριο. Ας τη διακόψουμε για τρίτη φορά, για λίγα λεπτά, μέχρι να καταφτάσει ο κύριος Ιακολίνο. Uh, Να συνεχίσουμε, συνάδελφοι, γιατί ο εισηγητής. εισηγητή. you Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2013 παρουσίασε την πρότασή της για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γνωστή και ως ΕΠΟ. Οι συζητήσει είναι εξελίξει στο Συμβούλιο και όταν θα ολοκληρωθεί το θέμα στη συζήτηση με τα κράτη-μέλη θα σταλεί στο Κοινοβούλιο για σύμφωνη γνώμη, γιατί δεν είναι διαδικασία συναπόφαση, είναι διαδικασία απλώ σύμφωνη γνώμη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιε επιφυλάξει σε κάποια κράτη-μέλη για την πρόταση. Εν ώψη λοιπόν τη σύμφωνης γνώμη, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών αποφάσισε να συντάξει μια ενδιάμεση έκθεση βάσει του κανόνα 81.3 για το πώ πρέπει να διαμορφωθεί η εισαγγελία και πώ θα πρέπει να ε, γίνει ώστε να λάβει και τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριο Ιακολίνο είναι ο εισηγητής, έλαβε 125 τροπολογίε και θα συζητήσουμε τι τροπολογίε σήμερα. Um, να ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κύριο Ιακολίνο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εξηγήσατε σαφέστατα από πού προέκυψε αυτή η πρόταση. Το Κοινοβούλιο μέσω μιας έκθεσης θα πρέπει να συνεισφέρει συγκεκριμένα. Κατατέθησαν 125 τροπολογίες, κάποιες από πλευράς μου, κάποιες άλλες από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Λίγο πολύ είναι μια όμορφη κατανομή και στόχος ε, είναι να τελειοποιήσουμε και να βελτιώσουμε ένα κείμενο το οποίο ε, στόχο έχει να μας κάνει να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα αυτή την ομοθεσία που ε, θα έχουμε μέχρι το τέλος της θητείας και να μπορέσουμε να εκφράσουμε ίσως και την άποψη του Κοινοβουλίου. Όπως θα γνωρίζετε για αυτό το προκαταρκτικό σχέδιο υπήρξε μια διαμάχη για την αρμοδιότητα με την Επιτροπή ε, ελέγχου του προϋπολογισμού ε, και η αρμοδιότητα αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο το προκαταρκτικό σχέδιο και όχι ε, το θέμα αυτό καθε αυτό. Αυτό όταν θα υποβληθεί η πρόταση θα πρέπει να εκφράσουμε την άποψή μας. εργάζονται επί του θέματος και άλλες επιτροπές και η Επιτροπή Κοντ, γι' αυτό ακριβώς και το χρονοδιάγραμμά μας έχει κάποιες μικρές αλλαγές για την ημέρα της ψηφοφορίας πιο συγκεκριμένα οριστικοποιήθηκε πλέον. Ε, θα ψηφίσουμε στις 20 Σεπτεμβρίου. Ε, θα περάσω στις διάφορες συνεισφορές που είχαμε και από τους κοιόδης συζητητές αλλά και πολλούς άλλους συναδέλφους οι οποίοι θέλησαν και αυτοί να εκφράσουν την υποστήριξή τους για ένα κείμενο το οποίο ε, σίγουρα χρειάζεται προσαρμογή και βελτίωση. Η συνάδελφος ε, Σίπελ ε, μας έκανε μια γενική παρατήρηση για κατανομή της συνεισφοράς μεταξύ γενικών υποδείξεων και νομοθετικών προτάσεων. Θα τα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα, θα τα συζητήσουμε και στους κοιόδης εισηγητές. Προβλέπεται συζήτηση στο Στρασβούργο στις 8 το πρωί και ελπίζω η προσέγγιση να είναι ισορροπημένη. Υπάρχουν επίσης κάποια... Ε, στοιχεία που αφορούν τις διάφορες απόψεις, παρά το γεγονός ότι η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι έτοιμη, αλλά τα υπόλοιπα θέματα θα τα ε, προσέξουμε ιδιαίτερα. Όσον αφορά τις αιτιολογικές σκέψεις, θα πρέπει να ε, συνεννοηθούμε όσον αφορά την προστιθέμενη αξία που θέλουμε να προσδώσουμε στο ρόλο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα ως ε, θεματοφύλακα των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνέπειες που υπάρχουν κυρίως στον προπολογισμό. Υπάρχουν αυτή η διαβόητη κίτρινη κάρτα η οποία ακόμα δεν ολοκληρώθηκε στο Συμβούλιο όπως τα γνωρίζετε. Ε, οι διαπραγματεύσεις είναι εν και κάθε άλλο παρά είναι και όπως είπε και η Πρόεδρος πριν από λίγο. Στην παράγραφο 1 υπάρχουν ε, κάποιες ε, πολύ συγκεκριμένε αναφορές ε, της συναδέλφου Κοράτσα Μπίλτ, την οποία βλέπω μεταξύ των παρισταμένων σε αυτή την ημέρα που είναι γεμάτη δουλειά για όλους μας και υπάρχουν και κάποιες παρεμβάσεις της συναδέλφου Σίπελ και της κυρίας Μακοβέη και της κυρίας Ματιέ. Και τα δύο θέματα της ενισχυσμένης συνεργασίας και της ομοφωνίας θα πρέπει να τα αναφέρουμε πολύ συγκεκριμένα και πολύ ισορροπημένα, διότι η διαδικασία είναι ακόμα εν εξελίξη, κυρίως το θέμα αυτή εδώ της κίτρινης κάθετας, όπως γνωρίζετε, ε, επισήμως δεν έχει ακόμα ε, συζητηθεί όπως προβλέπεται από το Συμβούλιο. Έχει ακουστεί βέβαια ότι θα γίνει, αλλά ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Έχουμε επίσης κάποιες προτάσεις για το επόμενο βήμα. Τα ε, διεθνή σοβαρά εγκλήματα. Υπάρχει και το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος. Εγώ ήμουν εισηγητή στην Ειδική Επιτροπή για το θέμα αυτό και νομίζω ότι ε, στο πρώτο ε, στάδιο θα πρέπει ε, η Ευρωπαϊκή Συγγελία να ασχοληθεί με αδικήματα που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια άλλη νομοθετική πρόταση για να εξετάσουμε και να καθορίσουμε σαφώς τις ε, αρμοδιότητες και τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι άλλως δεν θα υπήρχε λόγος να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Και επίσης μου φαίνονται λογικά τα όσα έχουν συνεισφέρει οι συνάδελφοι ε, στην παράγραφο 4 σημείο ε για τον ε, δικαστή και ε, στην επόμενη παράγραφη όμως το 4η θα πρέπει να υπάρχει αναφορά παρά το γεγονός ότι μπορεί και να υπονοείται απλώς στη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας για την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα συμπληρωματικά δικήματα και υπάρχει και το θέμα των οικονομικών συμφερόντων μεν, ε, θίγονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ε, αυτή θα είναι η φυσική αρμοδιότητα της εισαγγελία, αλλά υπάρχουν και πολλά παρελκόμενα σε αυτές τις περιπτώσεις και θα πρέπει να τα εξετάσουμε και αυτά. Όσον αφορά τις ε, δυνατότητες ανάκρισης και έρευνες, πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο forum shopping, το να επιλέξει κανείς δηλαδή το κατάλληλο δικαστήριο και υπάρχουν και κάποιες παράγραφοι που αφορούν θεωρούν το παραδεκτό των αποδείξεων ε, και η κυρία Σίπελ ε, μαζί με κάποια άλλα συνάδελφο ε, συνεισέφεραν και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε συμβιβασμό και ε, την αναφορά στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και στην παράγραφο αυτή έχουμε και μια συμβιβαστική λύση για την, τον ε, έλεγχο, το δικαστικό έλεγχο. Θα πρέπει όμως να αντιληφθούμε και να αποφασίσουμε ε, τι ποινές επιβάλλονται, για ποια δικήματα, για να ε, ε, μην είναι και ιδιαίτερα επιβαρημένη η δραστηριότητα του εισαγγελέα. Και επίσης υπάρχει και μια τροπολογία της κυρία Σίπελ που σχετίζεται με τον ε, δικαστικό έλεγχο και τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας στις οποίες αναφέρονται τα θέματα αυτά. Υπάρχουν κάποιες άλλες παράγραφοι που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψη και αθώς και άλλα θέματα που σχετίζονται με την νομιμοποίηση του ελέγχου και όλα αυτά θα τα λάβουμε υπόψη όταν θα ε, καθορίσουμε ποιες θα είναι οι συμβαστικές μας λύσεις. Επίσης, στις συμβαστικές προτάσεις θα πρέπει να δούμε ε, και τι γίνεται με τα δικαιώματα του κατηγορουμένου. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ε, προσέξουμε. Ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε, μην με κοιτάτε έξι. Η προστασία προσωπικών δεδομένων δεν προσπαθήσαμε να μην παραλείψουμε τίποτα και θα αναφερθούμε και σε αυτούν. Στα θέματα προστασίας δεδομένων έχουμε αρκετές τροπολογίες, θα προσπαθήσουμε και εδώ να βρούμε μια ισορροπία για να προχωρήσουμε. Η κυρία Βέμπερ αναφέρθηκε αρκετές φορές ε, και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αφορούν ε, τους, ε, τις διεθνείς οργανώσεις. Όσον αφορά τη φύση της ίδιας της αγγελίας, εμείς θέλουμε να είναι ένα ευέλικτο σχήμα και θεωρούμε ότι οι τροπολογίες οι οποίες επευλήθησαν θα είναι χρήσιμες για να εξετάσουμε το θέμα της αγγελίας. Αυτές είναι λοιπόν οι πρώτες μου παρατηρήσεις. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους και οδησυγητές, αλλά όχι μόνον αυτούς, διότι έδωσαν τις ε, παρατηρήσεις τους στη γραμματεία και σε μένα και ευχαριστώ ε, γιατί όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και θα ληφθούν δεόντως υπόψη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. you... Ευχαριστώ, λόγος που σας κοιτούσα έτσι. Είναι ότι έχουμε διακόψει τρεις φορές και μας μένουν μόνο 15 λεπτά. Τώρα, έχοντας διακόψει τρεις φορές δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα καταφέρουμε να, να, τελειώσουμε τη συνεδρίαση μετά από το καθορισμένο όριο. Εν πάση περιπτώσει, Αναγκάζομαι να περιορίσω το χρόνο ομιλία των υπολείπων ε, για την Επιτροπή και για το, την Ελληνική Προεδρία στα δύο λεπτά. Η Επιτροπή πρώτα και μετά η Προεδρία. Το μέγιστο δύο λεπτά παρακαλώ. Πριν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Χαιρόμαστε, καλωσορίζουμε την έκθεση του κυρίου Γιακολίνο και συμφωνούμε με την ουσία της. Πρόκειται για μια πρόταση στην οποία θα πρέπει να συμφωνήσει πρώτα το Συμβούλιο και έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσει. Μετά θα δοθεί η σχετική εντολή στην Επιτροπή. Τώρα έκαναν ορισμένε παρατηρήσει στα ε, μέλη του Κοινοβουλίου, αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την άποψη, τη θέση που θα λάβει το Συμβούλιο. Η διαδικασία συνεχίζεται, επομένω. Ευχαριστούμε. Η Ελληνική Προεδρία φαίνεται δεν εκπροσωπείται. Τέλο πάντων, αυτό μα δίνει λίγο περισσότερο χρόνο. Κυρία Σίπολ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας είναι νέος θεσμός. Νόημα έχει μόνο εάν μπορεί να πει κανείς ότι ο νέος αυτός θεσμός είναι αυτή η αρχή θα προσφέρει μια προστιθέμενη αξία απέναντι στην υπάρχουσα κατάσταση. Και η προστιθέμενη αυτή αξία δεν μπορεί παρά να έγκυται μόνο στην πραγματική δίωξη των εγκλημάτων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Όμως ή δυνατόν στη βάση ενιαίων κανόνων και σε ό,τι αφορά τους ουσιαστικούς και τους δικονομικούς κανόνες και εκείνους που προστατεύουν τα δικαιώματα των κατηγορουμένων, τα δικαιώματα προβολής ενστάσεων και εδώ η πρόταση της Κομισιόν μου φαίνεται κάπως να στερείται ισορροπίας διότι βλέπω ότι γίνονται πολλά πράγματα εθνικά. Εθνικά αρχίζει η δίωξη, εθνικοί κανόνες ισχύουν παρόλο που υπάρχει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Γι' αυτό εμείς εδώ έχουμε καταθέσει τροπολογίες για να επιτύχουμε ένα μέγιστο βαθμό εναρμονίσεως. Διότι αλλιώς πού βρίσκεται αυτή η προστιθέμενη αξία απέναντι στην νυν υφιστάμενη κατάσταση. Λέχθηκε επίσης ότι πρόκειται για διαδικασία σύμφωνης γνώμης. Άρα δεν μπορούμε να μπούμε σε όλα όπως σε συναπόφαση. Παρ' όλα αυτά η πολιτική μου ομάδα και εγώ αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε και συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις. Διότι θεωρούμε ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε διαδικασία σύμφωνης γνώμης φέρουμε την ευθύνη να πούμε με ακρίβεια ποια πορεία πρέπει να ακολουθήσει, ποιες είναι οι προσδοκίες μας. Και αυτό νομίζω ότι είναι και δίκαιο και έντιμο απέναντι στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο να πούμε τι ακριβώς θέλουμε, ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσει μας για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, έτσι ώστε πράγματι να μπορέσει να ασκήσει τα καθήκοντά του για προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και εν τέλει, στο κάτω γραφής, των συμφερόντων των δικαιωμάτων του φορολογουμένου. Ο εισηγητής τα εξήγησε ήδη στην εισαγωγή του. Δεν θα αρκεστούμε σε γενικές μόνο παρατηρήσεις για τα δίκαια του Ευρωπαίου Αγγελέου, δηλαδή για τις ε, αρμοδιότητές του. Θα κάνουμε και γενικότερες νομοθετικές προτάσεις. Ελπίζουμε να τα δεχθούν αυτά και οι άλλοι εισηγητέ, ώστε να διατυπωθεί μια εντελώς συγκεκριμένη πρόταση. Διότι επαναλαμβάνω ότι ο Ευρωπαίο Αγγελέας είναι καλή ιδέα, πρέπει όμως να μπορέσει να λειτουργήσει, πρέπει να προσφέρει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση. Και αντιμετωπίζουμε πάντοτε το πρόβλημα ότι δεν έχουμε λάβει αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα θέματα μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εκεί όπου έχουμε λάβει αποφάσεις για τον, για τον οδικό χάρτη, ακόμα αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν υιοθετηθεί στις χώρες μέλη. Και εδώ λοιπόν επισημαίνω ότι χρειαζόμαστε για να εξασφαλιστεί η προσθέμενη αξία του Ευρωπαίου Εισαγγελέως περισσότερη εναρμόνιση. Πάντως, τελευταία μου φράση αυτή, ακούστηκε ήδη σήμερα ότι χρειαζόμαστε βέβαια μια πολιτική των πολλών και μικρών βημάτων. Ευχαριστώ κυρία Βέμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως τα έχουμε ξαναπεί άλλες φορές και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ αλλά και στη συναντήση των σκιωδών εισηγητών θα ξαναπώ ότι η πρόταση είναι βέβαια ορθή κατά την πρόθεσή της αλλά απέχει πολύ από το να είναι καλή πρόταση όπως τουλάχιστον προτάθηκε στο Κοινοβούλιο. Εγώ επέμεινα ότι η πρόταση της Κομισιόν υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 86 και στερεί το Κοινοβούλιο από τα δικαιώματά του να συνομοθετήσει σε ό,τι αφορά την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και αυτή είναι και η γνώμη της νομικής μας υπηρεσίας. Όσον αφορά τις τροπολογίες, και βέβαια θα συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα και θα προσπαθήσουμε να, να δούμε, να συζητήσουμε, να εξετάσουμε τις συμβαστικές επιλογές και τη γραμμή των ψηφοφοριών. Όμως εγώ θα δεχθώ τις τροπολογίες Ζίπελ και Φως που προτείνουν ενισχυμένη συνεργασία. Και άρα η υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποβάλει νέα πρόταση. Νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος, ο σωστός δρόμος επί του παρόντος. Κατανοώ επίσης μάλλον μαθαίνω ότι και οι συνάδελφοί μας της Επιτροπής Προϋπολογισμών Υποβάλλουν τροπολογίες για να ζητήσουν από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να αναμείνει, να μην καταθέσει έκθεση πριν από τις εκλογές. Διότι έχω βέβαια κάθε σεβασμό για τους συναδέλφους μου της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, αλλά όταν εξετάζω τις τροπολογίες, τις ορισμένες εξ αυτών, καθίσταται σαφές για μένα ότι η ματιά που ρίχνουν είναι πολύ επιφανειακή. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι η πρόταση αυτή δεν συνοδεύεται από πρόταση για ευρωπαϊκό ποινικό δικαστήριο. Μα τι σχέση έχει. Και επίσης ζητούν να ε, θεσπιστούν και ειδικά κονδύλια για δικαστική αρρωγή ή για το ευεργέτημα παινίας ενώπιον των δικαστηρίων για πρόσωπα τα οποία διώκονται. Δεν καταλαβαίνω τι σχέση έχει. Έχουμε τελικά πρόταση για την χορήγηση του ευεργετήματος της παινίας. Βρίσκω λοιπόν αυτά τα πράγματα έχουν γίνει με ιδιαίτερη βιασύνη και δεν θα έπρεπε να τα δεχτούμε. Ευχαριστώ, ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανάπτυξη του θέματος και για τη δυνατότητα να σχολιάσουμε, έστω και σύντομα. Για το θέμα των προτύπων διαδικασίας θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Θα πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες για τις περιπτώσεις όπου μπορεί να προβεί σε έρευνες ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Πρέπει να εξασφαλιστεί και η νομική προστασία των θυγωμένων. Χρειάζεται λοιπόν να πούμε εμείς καθαρά τη γνώμη μας. Το ίδιο για την κρίση για τις αρμοδιότητες μέσα στην ίδια εισαγγελία που πρέπει να μπορεί να εξεταστεί και των, εκ των υστέρων. Εδώ χρειάζεται, χρειάζεται θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για να αποφευθούν ενδεχόμενα και ένα δικαίου στο τέλος. Επίσης θεωρώ ότι πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι τροποποιήσεις που θα εγκρίνουμε και εγώ είμαι διατεθειμένος να συνεργαστώ για να προκύψουν συμβαστικές τροπολογίες να ληφθούν σοβαρά υπόψη από το Συμβούλιο των Υπουργών. Και θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να εγκρίνουμε εν τέλει θέση η οποία θα περιλαμβάνει πολύ ξεκάθαρα ουσιαστικά στοιχεία και να έχουμε τη δυνατότητα μετά να επανέλθουμε, να παρέμβουμε ξανά στην παρατηνόμενη συζήτηση στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ τον Σαλβατόρη Ακολίνο για την καλή δουλειά που έκανε και την δέσμευση που ανέλαβε να ακούσει και να συμπεριλάβει τις γνώμες μας. Υπάρχουν 14 κοινοβούλια, εθνικό, εθνικά κοινοβούλια που ήγηραν την κίτρινη κάρτα της επικουρικότητας θα πρέπει η ε, Κομισιόν να υποβάλει νέα πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των Εθνικών Κοινοβουλίων, διότι αλλιώς υπονομεύουμε την ε, συνθήκη της Λισαβόνας και τη σχέση που έχουμε με τις Εθνικές Βουλές. Και ε, διερωτώνται οι πολίτες τι κάνει το Κοινοβούλιο με την επικουρικότητα. Έχω υποβάλει και τροπολογίες για την υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων, καθώς επίσης και για την προσφυγή κατά των αποφάσεων του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Διότι χρειαζόμαστε ασφάλεια δικαίου. Πρέπει να αποφευθούν οι εισδήποτε επικαλύψεις και να δούμε πού ακριβώς υπάρχουν οι συμβατότητες μεταξύ των διαφορετικών νομικών συστημάτων των χωρών μελών. Για παράδειγμα, οι έρευνες. Δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει το σύστημα που προτείνεται των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων. Νομίζω ότι η έρευνα θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Με λίγα λόγια, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και επομένως την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε τις απάτες κατά του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Δεν μπορούμε όμως να μπούμε τόσο πολύ μέσα στην επικουρικότητα και σε θέματα εθνικών ποινικών δικαίων. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε λοιπόν να αναθεωρήσουμε εντελώ το κείμενο, διότι αλλιώ θα είναι αδύνατον για μας να το υποστηρίξουμε. Then we come back to our for his concluding. Να επανέλθουμε στον συγητή λοιπόν για να ολοκληρώσει. Sì, ε, ε, Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή και την άποψη των σχεδόν εισηγητών την οποία σε κάποιο βαθμό γνώριζα άλλωστε, όπως για παράδειγμα την άποψη της κυρίας Κορατσαμπίλτ και την, κυρία, και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σαφές ότι αν δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία πολύ συγκεκριμένη για το θέμα αυτό, για τα ε, οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει κανένα νόημα. Η κοινή προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε λοιπόν εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να εκφράσουμε ίσως και μια επίκριση ε, ενώπιον των επιλογών ε, που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή το να δρανίσουμε και να δώσουμε ένα σαφή προσανατολισμό από πλευράς Κοινοβουλίου κατά με είναι πολύ ξεκάθαρο. Πάντα πρέπει να εκφράζουμε τουλάχιστον την άποψή μας. Πρέπει να την εκφράζουμε τουλάχιστον γνωρίζοντας ότι ο ρόλος μας είναι συγκεκριμένο και είναι αυτό το οποίο έχουμε αναλάβει να κάνουμε. Σαφώς και οι άλλες επιτροπές θα μπορέσουν να συνεισφέρουν και αυτές με τη σειρά τους. Τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών σίγουρα ενδιαφέρονται για έναν οργανισμό ο οποίος θα έχει σαφείς και καθορισμένες αρμοδιότητες, που θα υπάρχει ένας αρχικός δικαστής ε, που θα έχει συγκεκριμένα δικαιώματα. Αν όλα αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε σε ένα προκαταρκτικό σχέδιο, το οποίο δεν αποκλείει το γεγονός να υπάρξουν και άλλα μέχρι το Συμβούλιο να καταθέσει μια πρόταση που ίσως να λάβει υπόψη και του προσανατολισμού μας. Εμείς δεν έχουμε καμία δυνατότητα εδώ να ε, να συνεισφέρουμε ούτε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε ως ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε προς το Συμβούλιο. Εμείς απλώς θα πρέπει να δώσουμε μια άποψη με σαφείς υποδείξεις ε, για το τι ακριβώς θέλουμε, για να έχουμε μια δομή η οποία θα είναι ευέλικτη και σύγχρονη και θα μπορέσει να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε καταλήλως τους κοινοτικού πόρους. Αυτή είναι η προσδοκία μας και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και για την ενισχυμένη συνεργασία θα το δούμε το θέμα αυτό και τις επόμενες ημέρες και ώρες με τους κοιόδης συγητές για να δούμε ποια είναι η πιο συνεκτική λύση για όλα όσα έχει πει ο καθένας μέχρι τώρα με πάσα ειλικρίνεια, με πάσα ερεμία προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε μια δομή που θα πρέπει, όπως είπαν και άλλοι, το επαναλαμβάνω και εγώ, να δώσει μια προστιθέμενη αξία για την κατάλληλη χρήση όλων των ευρωπαϊκών πόρων ώστε να έχουμε καλύτερη ευημερία, καλύτερο πολιτισμό, μια καλύτερη προσέγγιση ενώπιον της μετανάστευσης και ε, να μπορούμε να βοηθήσουμε και τα πανεπιστήμια και την έρευνα. Και όλα αυτά είναι πόροι οι οποίοι θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι τόσο σημαντική. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της συνεδρίασης για σήμερα το πρωί. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι σήμερα το απόγευμα η συνεδρία είναι στην αίθουσα 3 σε 50 στο άλλο κτίριο και επίσης να σας ενημερώσω ότι σήμερα το απόγευμα εάν πάλι ε, προχωράμε πιο γρήγορα. Δεν θα κάνω αναβολή επί αναβολή. Σας παρακαλώ όλους να είστε λίγο πιο έγκαιρα στην ώρα σα για τα θέματα τη μέρας τη διάταξης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, γιατί πραγματικά δεν είναι δυνατόν να διακόπτουμε συνέχεια για μισή ώρα. Αν δεν υπάρχουν αρκετά μέλη, το καλύτερο θα ήταν να ε, ολοκληρώσουμε με την ημερήσια διάταξη και να φύγουμε νωρίτερα και όχι να διακόπτουμε συνεχώς. Τα λέμε το απόγευμα.